Mes Ας ξεκινήσουμε αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαστε στην αίθουσα συνεδριάσεων της ομάδας του ΕΛΚ, την παλιά αίθουσα συνεδριάσεων της αίθουσας της, ε, του ΕΛΚ. Εδώ παλιά, μια φορά και έναν καιρό, συνεδρίαζε η συνέλευση για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη απουσία μελών εκτός από τον ε, συνάδελφο Ναραχό τον οποίο χαιρετώ διότι το ΕΛΚ έχει το συνεδριό του σήμερα και αύριο στο Βουκουρέστι και επομένως μερικοί μοναχα από εμάς έχουμε μείνει εδώ ως όμοιροι. Λοιπόν, πρέπει να δούμε αν έχουμε απαρτία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες βέβαια με την πολιτική ισορροπία που ισχύει σήμερα. Ξέρετε ότι αρχικά είχαμε προβλέψει να συνεδριάσουμε όλη μέρα αλλά συμφωνήσαμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα θέματα και να κάνουμε και τις ψηφοφορίες το πρωί. Και έτσι θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε ένα αρκετά ταχύ ρυθμό για να μπορέσουμε να διεκπαιρεώσουμε όλα αυτά τα θέματα. Είδατε την ημερήσια διάταξη. Δεν υπάρχουν ε, παρατηρήσεις για την ημερήσια διάταξη, οπότε μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει εγκριθεί. Οι παρατηρήσεις του Προέδρου βρίσκονται στο έγκριτο έντυπο κόμπου News. ανακοινώνεται ένα σεμινάριο στις 7 Νοεμβρίου με δημοσιογράφους με θέμα το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σημείο 3. Εδώ πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά της συνεδριάσεώς μας της 8 Οκτωβρίου. Πώς ήθιστε, εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι το τέλος της συνεδρίας, θα θεωρήσουμε ότι τα πρακτικά αυτά έχουν εγκριθεί. τριμέρες διάλογος για τον προϋπολογισμό που έλαβε χώρα χθες. Ο εισηγητής μας, ο Τζοβάνι Λαβία, δυστυχώς δεν μπορεί να είναι παρόν. Βρίσκεται μακριά μακριά και έχει και να διεξαγάγει προεκλογική εξαρτία στη Σικελία. Μπορώ να κάνω ίσως μια παρουσίαση σύντομη και ίσως η Ιούτα και ο Δέρεκ Βόαν μπορούν να συμπληρώσουν αυτά τα οποία θα πω. Ο τρίλογος αυτός ήταν τυπικού χαρακτήρα. Ως αντικείμενο είχε τον προϋπολογισμό του 2013 και παρουσίασαν οι συγητές μας τις προτεραιότητες για τις οποίες έχει συμφωνήσει και ψηφίσει η Επιτροπή Προϋπολογισμού και τις οποίες θα παρουσιάσουμε στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα. Έλαβε χώρα και μια ανταλλαγή απόψεων για τους αποκεντρωμένους φορείς. Είναι τρεις οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται με την εφαρμογή του άρθρου 47 της ε, Διαθεσμικής Διοργανικής ε, Συμφωνίας. Εμείς προτείναμε μαζί με την Κομισιόν να υπάρξει μια κοινή δήλωση των τριών θεσμικών, βασικών θεσμικών οργάνων για τους αποκεντρωμένους φορείς. Το Συμβούλιο είπε ότι δεν είναι εχθρικό προς μια τέτοια συμφωνία, αλλά δεν ήταν ακόμα έτοιμο να συμφωνήσει. αλλά νομίζω ότι τελικά θα συμφωνήσει. Επίσης, συζητήσαμε για το πρόβλημα των πιστώσεων πληρωμών, το πρόβλημα συμπληρωματικών πληρωμών που χρειάζονται. Η Φρανσιάσκα Μπαλτσάν είναι εδώ και δεν μπορεί να αναφερθεί στα θέματα αυτά. Από το 2012 ήδη θα χρειαστούμε ήδη από τώρα, δηλαδή θα χρειαστούμε κάποιες πιστώσεις πληρωμών και πρέπει να αξιολογήσουμε και τις ανάγκες για το 2013 από την πλευρά του Κοινοβουλίου. Αποφασίσαμε με τους συντονιστές ότι μπορούμε να κάνουμε μια συγκεκριμένη πρόταση σε σχέση με τη μέθοδο που θα πρέπει να ακολουθηθεί ή καλύτερα για την αλλαγή της μεθόδου που πρέπει να ακολουθηθεί προς το Συμβουλίο και την Κομισιόν για την, για την εκτίμηση των ε, πιστώσεων πληρωμών. Έχω διανύμει σε εσάς ένα μη έγγραφο που προέκυψε μετά από τη συνάντηση, την τριμερή συνάντηση που κάναμε πριν από τρεις εβδομάδες μαζί με τον Επίτροπο Λεβεντόφσκι και τον Υπουργό Μαυρογιάννη από την Κυπριακή Προεδρία, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα με ποιο τρόπο γινόταν η αξιολόγηση των πιστώσεων πληρωμών μέχρι τώρα, γιατί πολλές φορές καταλήγαμε σε παρεξήγηση μεταξύ των τριών μεγάλων θεσμικών οργάνων και πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή την τόσο δυσάρεστη κατάσταση. Θεωρήσαμε λοιπόν με την ευκαιρία αυτής της συνάντησης του τριμερούς διαλόγου πριν από τρει εβδομάδε, ότι η τωρινή διαδικασία η οποία επιτρέπει στην Κομισιόν να <clears throat> προβαίνει σε μία αξιολόγηση και να μας προτείνει συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία ήταν πολυδέδαλη, σκοτεινή και οδηγούσε σε παρεξηγήσεις. Ο στόχος μας, και το λέω σαφώς, και προς το Συμβούλιο, είναι να επανέλθουμε σε μία κατάσταση που θα έπρεπε να είχε παραμείνει ούτως, βάσει της οποίας η πολιτική διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό σε αιτήσιο επίπεδο και, οι και τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς γίνεται πρώτα για τις πιστώσεις υποχρεώσεων και στη συνέχεια ακολουθεί η συζήτηση για τις ε, πιστώσεις πυλωμών σε τεχνικό επίπεδο και δεν πρέπει να εμπλακεί η πολιτική συζήτηση παρά μόνο αν υπάρχουν απρόοπτα. Ο τρόπος για να μπορέσουμε να επιτύχουμε κάτι τέτοιο όπως, προτεν, όπως αναφέρουμε στο μη γραφό μας είναι να προσκαλέσουμε κάθε κράτος μέλος να συγκεντρώσει σε ένα κεντρικό φορέα λογικά θα είναι το Υπουργείο Οικονομίας ή Εθνικής Οικονομίας αλλά κάθε χώρα πρέπει να αποφασίσει μόνη της να συγκεντρώσει τις ε, εκτιμήσεις για, ανα, για ανάγκες πιστός και τις αιτήσει επιστροφών που προς το παρόν παραμένουν στην ευθύνη των εθνικών διοικήσεων που διαχείριζονται τα εθνικά προγράμματα, των εθνικών ή υποεθνικών διοικήσεων και που αναφέρονται στην, ε, στους ομόλογούς τους στην Επιτροπή την αντίστοιχη Γενική Διεύθυνση δηλαδή της Κομισιόν και συνέχεια όλες οι Γενικές διευθύνσει τη Κομισιόν διαβιβάζουν με κάποιες προσαρμογές ενδεχομένως στην Γενική Διεύθυνση προπολογισμού τα στοιχεία αυτά. Αυτό το σύστημα είναι αδιαφανές, οδηγεί ορισμένες διοικήσεις στο να υπερεκτιμούν τι ανάγκε του και καταλήγει στο ότι παρά τις ε, οριζόντιες περικοπές που εφαρμόζει η Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού για τις αιτήσει αυτές, οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα το οποίο αναγκάζει τους Υπουργούς Οικονομικών να ολολίζουν στις συνεδριάσεις τους όταν βλέπουν τα αριθμητικά αυτά στοιχεία. Μετά από όλα αυτά, η πρόταση την οποία κάνουμε στοχεύει όχι να εμποδίσει, αλλά να βοηθήσει τους Υπουργούς προϋπολογισμού, προϋπολογισμών να αντιμετωπίσουν καλύτερα τα προβλήματα αυτά. Από τη στιγμή που η κάθε χώρα, και ξεκινώ από τη δική μου, έχει ένα, μια συγκέντρωση όλων των αιτήσεων στο Υπουργείο Οικονομικών για την εκτίμηση των αναγκών και των επιστροφών. Τότε το Υπουργείο αυτό θα τις πιστοποιήσει, θα τις δημοσιεύσει και έτσι θα μπορεί να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου εάν τα εθνικά ελεγκτικά όργανα θέλουν να προβούν σε ένα τέτοιο έλεγχο και στη συνέχεια θα στείλει τα στοιχεία αυτή, αυτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδανικά σε τέτοιες συνθήκες ώστε η Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού θα πρέπει μονάχα να κάνει μία πρόσθεση για τα στοιχεία που έρχονται από τις 27 χώρες και έτσι να γνωρίζει ποιες θα είναι οι πιστώσεις πληρωμών ως άθροισμα των 27 χωρών μελών που έχουν προτείνει Υπουργοί Οικονομικών, οι οποίοι στη συνέχεια δεν μπορούν να αντιταχθούν σε αυτά τα στοιχεία. Αν οι Υπουργοί τώρα Οικονομικών θεωρούν ότι το άθροισμα δεν είναι ορθό, αυτό θα πρέπει να το βρουν μεταξύ τους. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν πρέπει να εμπλέκει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να χρειάζεται να εκφέρει γνώμη σε σχέση με την αξιολόγηση, με την εκτίμηση των αναγκών όπως διατυπώνεται από τις αρχές διαχείρισης. Η Κομισιόν για τα προγράμματα που έχουν άμεση διαχείριση και εθνικές διαχείρισεις, εθνικές μάλλον διοικήσεις για τα προγράμματα με κοινή διαχείριση, θα πρέπει να αναλαμβάνουν τη διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των συναφών χρηματοδοτήσεων. Εμείς δεν έχουμε κανένα ρόλο σε αυτή την ε, διαχείριση. Ήδη έχουμε αρκετά προβλήματα με τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν και έχουμε ένα θαυμάσιο εισηγητή. Και δεν μπορεί κανείς να μας περιμένει, να περιμένει από εμά να διαμεσολαβούμε μεταξύ των διαφορετικών εκτιμήσεων της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να θεσπίσουμε ένα μηχανισμό τιούτων, ώστε τα προβλήματα των πληρωμών <clears throat> μπορούν να ρυθμίζονται μέσα σε ένα τεχνικό πλαίσιο. Και μόνο εάν τώρα που είμαστε στο τέλος περίοδου προγραμματισμού αναφιούν ανάγκες αντικειμενικές για χρηματοδότηση και ξέρουμε ότι και τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν πολλές φορές δυσκολίες για να τροφοδοτήσουν τον κοινωτικό προϋπολογισμό, τότε το θέμα αυτό μπορεί να συζητηθεί από τους αρμόδιους υπουργούς μαζί με την Κομισιόν και η δική μας παρέμβαση θα παραμείνει περιορισμένη. Τούτων λεχθέντο λοιπόν, εμείς έχουμε διατυπώσει αυτή την πρόταση. Δεν ξέρουμε κατά πόσο <clears throat> θα μπορέσει να εφαρμοστεί από τον διορθωτικό προϋπολογισμό του 2012, από τον τελευταίο διορθωτικό προϋπολογισμό του 2012 αλλά μας φαίνεται μια ενδιαφέρουσα ιδέα και αν επιτύχουμε μια συμφωνία στον επόμενο τριμερή διάλογο στη συνδιαλλαγή, τότε θα προτείνουμε να ενσωματωθεί στη διαθεσμική συμφωνία. Για τον διορθωτικό λοιπόν προϋπολογισμό του 2012, ξέρετε ότι είχαμε αναφερθεί την προηγούμενη εβδομάδα στον προϋπολογισμό υπαριθμών 5 και σήμερα θα ψηφίσουμε για αυτόν τον προϋπολογισμό. Έναντι του Συμβουλίου λοιπόν, κάναμε μια σαφή διάκριση μεταξύ του προϋπολογισμού υπαριθμών 5, του διορθωτικού 5 και του διορθωτικού 6. Ο 5 αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης σε σχέση με την περιφέρεια της Εμίλια Ρωμάνια που αντιμετώπισε σοβαρές κλιματικές συνθήκες και καταστροφές. Έχουμε ζητήσει τα θύματα αυτής της καταστροφής να μην αποβούν θύματα των εσωτερικών προβλημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολιτικό ή διοικητικό επίπεδο και να μην καθυστερήσουν οι αρρωγές και οι αποζημιώσεις τις οποίες χρειάζονται. Υπενθυμίσαμε επίσης ότι εάν το Συμβούλιο θεωρεί ότι βάσει του πρωτοκόλου υπαριθμών 1 της συνθήκης της Λισαβόνας χρειάζεται την άποψη των Εθνικών Κοινοβουλίων προτού να ψηφίσει σε σχέση με ένα σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού. Υπενθυμίζω ότι το ίδιο αυτό πρωτόκολλο προβλέπει τη δυνατότητα κατεπίγουσας δράσης που παρακάμπτει αυτή την ανάγκη διαβούλευσης όταν το απαιτούν οι συνθήκες και φυσικά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κατεπήγοντος όπως το τόνισε και ο πρόεδρος του Συμβουλίου και επιμείναμε δηλαδή για αυτό το λόγο ο διορθωτικός προϋπολογισμός υπαριθμών 5 να αντιμετωπιστεί χωριστά πριν από τον 6 και να μην αντιμετωπιστεί στην συνολική διαπραγμάτευση της συνολικής δέσμης για τον προϋπολογισμό του 2013 που έχει να κάνει με τον διορθωτικό προϋπολογισμό. Ο υπαριθμόν 6 τώρα. Εδώ μας κατάει σε αγωνία η Κομισιόν. Θα επιτρέψει αυτός ο διορθωτικός προπολογισμό να αντιμετωπίσουμε πιστώσει πληρωμών του 2012 που ξέρουμε ότι δεν είναι επαρκή κατά ένα μονοψήφιο αριθμό δισεκατομμυρίων, ενδεχομένω ένα διψήφιο αριθμό δισεκατομμυρίων. Αλλά η Κομισιόν δεν θα εγκρίνει αυτόν τον διορθωτικό προϋπολογισμό παρά στη συνεδρίασή της της επόμενης εβδομάδος. Μπορούμε να επανέλθουμε λοιπόν και είναι σαφές ότι όπως και τα, επόμενα, τα προηγούμενα χρόνια αυτός ο διορθωτικός προϋπολογισμός, η συζήτησή του θα συνδυαστεί με τη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2013. Φραντσέσκα, θέλεις να πεις κάτι? Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η εισαγωγή σας ήταν λεπτομερεστάτη και πλήρης. Νομίζω ότι μετά από τον τριμερή διάλογο που έγινε χθες θα ήταν καλό να συμπληρώσουμε την έκθεση για το συμπληρωματικό 5 σχετικά με τον κίνδυνο στον οποίο αναφερθήκατε την εφαρμογή του πρώτου πρωτοκόλου που δεν καλύπτεται αυτή τη στιγμή μόνο με μία τροπολογία, αλλά είναι κάτι το οποίο θα μπορέσει να μας παρασύρει, θα έλεγα, στη συναπόφαση που δεν είναι ο καταλληλότερος χώρος για μας για τη συζήτηση του Ταμείου Αλληλεγγύης. Προτείνω λοιπόν όταν περάσουμε στην ψηφοφορία για τον συμπληρωματικό 5 να εισάγουμε δύο νέες παραγράφους στην τροπολογία μου που διευκρινίζει ακριβώς την θέση του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής μας μάλλον, γύρω από την προβληματική αυτή. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Αυτή η προφορική τροπολογία θα είναι διαθέσιμη γραπτά. Προφορική γραπτά. Και θα την έχετε στη διάθεσή σας πριν από την ψηφοφορία. Ο Τέρεκ. Σύντομα θα είμαι, Πρόεδρε. Πράγματι με τους τριμερούς διαλόγους έχουμε την δυνατότητα να προωθήσουμε τις απόψεις του Κοινοβουλίου και στον τομέα του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου και σε σχέση με θέματα άλλα όπως το ίτερ κτλ. Η Επιτροπή αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχουμε κάνει για κάποιες έστω και μικρές αυξήσεις για τον επόμενο χρόνο. Όλοι έκαναν προσπάθειες βέβαια και τα άλλα όργανα έτσι ώστε να μείνουν όλες οι προτινόμενες αυξήσεις κάτω του 1,9% εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. Ελπίζω λοιπόν να γίνει δεκτή η πρόταση για το συμπληρωματικό προϋπολογισμό. Σχετικά τώρα με τον γενικό προϋπολογισμό, αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση ότι δύσκολα μπορεί να δεχθεί κανείς τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι σαν να μην πιστεύουν, θα έλεγα, τις καλές προθέσεις αυτοί που τις αμφισβητούν, που αμφισβητούν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βλέπουν τα θέματα με πάρα πολύ πολιτικό τρόπο και είναι πολύ δύσκολο να πείσουμε το Συμβούλιο να αλλάξει απόψεις και γι' αυτό νομίζω ότι θα παραταθούν όσο γίνεται αυτές οι συζητήσεις. Πολύ σύντομα. Τόσου πολλού τριμερεί διαλόγου που έχω κάνει, τόσε πολλέ ε, συνδιαλλαγές, δεν περίμενα το Συμβούλιο να μπορέσει να με κοροϊδέψει για άλλη μια φορά ή να με ξαφνιάσει καλύτερα. Πλην όμω, έχουμε την ε, μέθοδο που θέλαμε να ολοκληρώσουμε βάσει το άρθρο 27 και να κάνουμε και τη σχετική δήλωση. Ωστόσο, ούτε για τον προπολογισμό ούτε για το προσωπικό δεν υπήρχαν δυσκολίες και δεν έχουν συνέπειες αυτά τα μέτρα στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Το πρόσθετο δηλαδή προσωπικό που θα χρειαστεί θα ε, χρηματοδοτείται από τα τέλη. Ωστόσο το Συμβούλιο δεν είναι σε θέση να πει το ναι. Και αυτό πραγματικά με ξαφνιάζει. Εγώ περίμενα ότι θα ήταν αυτό το πιο αυτονόητο, το λιγότερο διαφιλονικούμενο από τα θέματα που είχαμε χτε να συζητήσουμε, αλλά το αναβάλει για άλλη μια φορά, που θα είχε μάλλον να συζητήσει, αλλά το αναβάλει για άλλη μια φορά το Συμβούλιο. Α περιμένουμε λοιπόν και α δούμε πού θα καταλήξουμε. Πάντω μου φαίνεται παράξενο. Και ώρες-ώρες έχω και την εντύπωση ότι αυτοί οι τριμερείς διάλογοι είναι μάλλον χάσιμο χρόνο. Ναι, έχει πάρει το χαρακτήρα τελετουργικού, σχεδόν ε, θρησκευτικού χαρακτήρα, λέει ο κύριος Λαμασούρα, απλώς δεν ξέρουμε ποιον Θεό πιστεύουμε. Λοιπόν, θα τελειώσουμε με μια γραπτή διαδικασία. Θα ήταν προτιμότερο αλλά πρέπει να κοιτάξουμε αυτό το κείμενο, το οποίο είναι πολύ σύντομα βεβαίω, που λέει και η Γιούτα ότι δεν υπάρχει λόγο ε, να υπάρχουν προβλήματα οικονομικού τύπου, διότι τα χρήματα δεν επιβαρύνουν τον ευρωπαϊκό, η χρηματοδότηση δεν επιβαρύνει τον ε, ευρωπαϊκό προπολογισμό. Και μετά κοιτάμε την παραδοσιακή διαδικασία. Προφανώ θα πρέπει να μεταφραστεί σε όλε τι ε, γλώσσε πριν να δοθεί η άδεια στον πρόεδρο του Συμβουλίου, το πράσινο φω δηλαδή από πλευρά του Συμβουλίου. Αυτά θα έχουμε πιστεύω σύντομα την γραπτή επιβεβαίωση από πλευρά του George Lyon τώρα. Πρόεδρε, ένα σχόλιο για τον on paper και ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν στον τριμήρη διάλογο για τη χάλη της μέρας Όταν μίλησε ο Ντέρεκ, νομίζω ότι στάθηκε σε θέματα που δεν έχουν τόσο πολύ ουσιαστικό χαρακτήρα, αλλά το θέμα δεν είναι τεχνικό. Είναι πολιτική απόφαση ότι δεν θέλει το 6,8 αύξηση στις πληρωμές του Συμβούλιο. Και τα δικά τους ε, νούμερα υποδεικνύουν τι περιμένουν από την επόμενη χρονιά. Εν πάση περιπτώσει, πολιτικά μπορεί κανείς να το χαρακτηρίσει είτε κοινική στάση είτε οτιδήποτε άλλο, αλλά επιμένουν στους δικούς τους, ε, στα δικά τους αριθμητικά. Και άρα το ζητούμενο για το Κοινοβούλιο είναι αν είναι διατεθειμένο να αγωνιστεί για την χρηματοδότηση που χρειαζόμαστε για τα ε, προγράμματα αυτά. Αλλά τα προγράμματα αυτά θα είναι ως όφελος των κρατών. επομένω, γιατί εμείς να αγωνιστούμε για κάτι το οποίο αφορά τα ίδια τα κράτη. Ο κύριος Λαμασού. Άκου να σου πω, Τζόρτζ. Οι υπουργοί του προπολογισμού των δημοσιονομικών στις περισσότερες χώρες δεν γνωρίζουν τι είδους ε, πιστώσεις πληρωμών αναλαμβάνουν οι άλλες διοικητικές μονάδες ή διοικητικοί φορεί των κρατών. Άρα, σε μια κεντρική δομή θα υπάρχει δυνατότητα για τον κάθε Υπουργό Δημόσιων Οικονομικών να ελέγχει, να αστυνομεύει την ίδια του τη χώρα. Ενδεχομένως δε και να περιστήλει προκαταβολικά τα αιτήματα για πιστώσεις πληρωμών του κάθε κράτος στις Βρυξέλλες, προς τις Βρυξέλλες. Εάν λοιπόν φανεί ότι παρά αυτή η προσπάθεια της αστυνόμευσης και της λιτότητας, στην οποία θα αποδηθούν όλοι οι υπουργοί των δημοσιονομικών στα κράτη, φανεί ότι τα 27 σύνολα ε, καταλήγουν σε, σε ποσό υψηλότερο από αυτό το οποίο θα μπορούσαν να, να θεωρηθούν ανεκτό οι υπουργοί στο Συμβούλιο, τότε η μπάλα θα είναι στο πεδίο των υπουργών αυτών τη εθνική οικονομία. Δηλαδή θα υποχρεωθούν εκείνοι να βρουν τι λύσει να περικόψουν προγράμματα ανακράτω σε κάθε περίπτωση. Άρα πρέπει να αναπέμψουμε σε αυτού τα θέματα που ανήκουν στι δικέ του αρμοδιότητε. Ίσως αυτό να είναι δύσκολο για τον προϋπολογισμό 2013 να το καταφέρουμε, να το εφαρμόσουμε. Αλλά και δεν ξέρω αν θα, είχε κάποιο, θα υπήρχε κάποια δυνατότητα για τον διορθωτικό προπολογισμό 2012 που σε μερικέ μέρε μόνο θα υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλλον θα είναι δυνατόν. Αλλά το σύστημα αυτό, τη, μηχανική αυτή λύση μπορούμε να την αξιοποιήσουμε για το μέλλον. Και θα δούμε πρακτικά τι ε, μα λένε και οι υπηρεσίε τη Επιτροπή αλλά και το Συμβούλιο. Ο κύριος Γκοτμάνη έχει. Ευχαριστώ πολύ. Δύο πράγματα. Remember in another trilogue. Ασχολούμαι και με το θέμα του Ταμείου Συνοχής όπου υπάρχουν αρκετά χρήματα αλλά και εκεί έχουμε συναντηθεί τέσσερις φορές και ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν έχουμε καταλήξει σε κανένα συμβιβαστικό σε αυτή τη φάση τουλάχιστον πεδίο. Από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να ετοιμαστούμε για συνδιαλλαγή. Δεν νομίζω ότι οι 10 ή 11 συναντήσεις τριμερούς επίπεδου θα οδηγήσουν πουθενά. Εμείς δεν θέλουμε να φτιάξουμε μια απλή γέφυρα από τον ένα στον άλλο προϋπολογισμό. Υποστηρίζουμε όμως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή μόνη της γνωρίζει τις οικονομικές μας υποχρεώσεις, τις νομικές μας υποχρεώσεις, τα περιθώρια, τα ανώτατα όρια, τα γνωρίζει και τα ελέγχει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν είναι το θέμα να χωριστούμε ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι πληρώνουν και σε αυτούς οι οποίοι δεν πληρώνουν. Νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να κάνουμε προτάσεις έτσι ώστε να μην χρειαστεί να αλλάξουμε το σύνολο του MFF. Είναι ο τελευταίος χρόνος με τον τρόπο αυτό που φτιάχνουμε προϋπολογισμούς. Αν τυχόν δεν κλείσουμε σωστά τον προϋπολογισμό, σαν παράδειγμα στο 1α, θα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Υπάρχει ας πούμε το θέμα των 50 εκατομμυρίων για την ευελιξία. Εκεί βέβαια τίθεται το θέμα. Σε άλλους τομείς ε, δεν τίθεται το θέμα. Αν θέλει το Συμβούλιο μειώσεις είναι κάτι το καινοτόμο ουσιαστικά. Ναι μεν θέλει να περικόψει το Συμβούλιο, θέλει να περικόψει συνολικά 5 δις, αλλά γιατί κάνετε τις περικοπές με αυτόν τον τρόπο πρέπει να τους ρωτήσουμε και με όχι με άλλο τρόπο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για την επόμενη συνάντηση κορυφής. Κατανοούμε ότι δεν μπορούμε να μεγαλώνουμε τους προϋπολογισμούς. Το θέμα είναι να κλείσουμε τους προϋπολογισμούς. Αν δεν κλείσουμε τακτικά τον προϋπολογισμό αυτόν τον οποίο τρέχουμε τώρα, ε, θα έχουμε προβλήματα. Θα στείλουν την Επιτροπή, θα παρέμβει το δικαστήριο, ο Λεβαντόφσκι τα έχει πει αυτά πάρα πολύ καλά. Θα λείπουν εκατομμύρια για το Εράσμους, θα δημιουργηθούν πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, αν μας τριμώξουν τόσο πολύ όσο μας τρίμωξαν τα τελευταία δύο χρόνια και στις πληρωμές και δυστυχώς μπορεί να έχουν την δυνατότητα αυτή, δεν ξέρω πόσο σοβαρές είναι οι προθέσεις τους, αν καταλήξουν μεταξύ τους σε μια κάποια συμφωνία, τότε εμείς καλούμεθα να διαχειριστούμε τις συνέπειες. Αν εμείς σταθούμε όμως μόνο στη διαχείριση των αρνητικών αποτελεσμάτων, τα πράγματα για μας θα είναι πολύ άσχημα. Ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό λοιπόν και θα σας πρότεινα εξάλλου να περάσουμε στο σημείο 4 λέω πρώτος της ημερησίας διάταξης συνεχίζοντας αυτά που είπαμε ναι, θα επανέλθουμε στο σημείο 6 για, τον, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού υπαριθμών 5 που θα ψηφίσουμε τώρα αλλά επειδή ήδη αναφερόμαστε στον προϋπολογισμό αυτό και στον προϋπολογισμό του επομένου έτους να μας παρουσιάσει τη θέση της η Φραντσέσκα με την προφορική της τροπολογία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχουμε ήδη εν πολλής ασχοληθεί με τον πέμπτο συμπληρωματικό, διορθωτικό. Συνδέεται με το θέμα των πληρωμών και του τριμερούς διαλόγου που έγινε χθε. Τα πιο σημαντικά σημεία τα είπατε η ατυχής επιθυμία του Συμβουλίου να θεωρήσει ότι εφαρμόζονται οι οκτώ εβδομάδες για την διαβούλευση με τα κοινοβούλια στα πλαίσια του πρωτοκόλου 1. Κάτι τέτοιο θα μας ε, οδηγήσει σε παράταση δύο μηνών της διαδικασίας και θα μας οδηγήσει τελικά με το ζόρι στην ε, συνδιαλλαγή για τον προϋπολογισμό του 2013. Γι' αυτό και προτείνω την προφορική τροπολογία, την οποία έχετε λάβει γραπτά, που εισάγει δύο νέες παραγράφους στο εσωτερικό του αρχικού κειμένου. Υπογραμμίζουμε την δεδηλωμένη πεποίθηση του Συμβουλίου ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει δύο επιπλέον εβδομάδες και αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας οδηγήσει το πέρασμα, το υποχρεωτικό του διορθωτικού 5 στη συνδιαλλαγή. Κανονικά θα έπρεπε επίσης να ψηφίσουμε τον συμπληρωματικό 5 ακόμα και σήμερα, χωρίς να έχουμε τη θέση την τελική του Συμβουλίου, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια τελική θέση στην Ολομέλεια τον μήνα Νοέμβριο και να κλείσουμε έτσι τη διαδικασία της διαμόρφωσης της κοινοβουλευτικής άποψης. Αν θέλουμε να κρατήσουμε αυτή τη στρατηγική επιλογή που είναι η καλύτερη, θα πρέπει να υπερψηφίσουμε σήμερα μέσω της τροπολογίας και όλας και τον διορθωτικό 5. Αυτές είναι οι μοναδικές άλλωστε τροπολογίες στο έγγραφο που έχουμε ήδη συζητήσει. Η προθεσμία της 15ης Οκτωβρίου που είχε υπάρξει για τις τροπολογίες δεν είδε να κατατίθενται νέες προτάσεις και μόνο υπάρχει ουσιαστικά η προφορική τροπολογία με τις δύο νέες παραγράφους. Λοιπόν, χωρίς να έχει άποψη ακόμα εκφράσει το Συμβούλιο, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη διαδικασία τη δική μας τον Νοέμβριο, να υπερψηφίσουμε την πρόταση σήμερα, συμπληρωματικά. Θα πρέπει να ψηφίσουμε επίσης και τη νομική βάση για την χρήση του Ταμείου. Ο εισηγητής μας είναι όμως το Βουκουρέστι με το ΕΛΚ και μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω. Σύντομα θα πω το εξής. Έχετε καταρχάς τις πληροφορίες που απαιτούνται στα πλαίσια του Com News. Θα πρέπει να βοηθήσουμε την περιοχή της Εμίλια Ρωμάνια που χτυπήθηκε από επανειλημμένους σεισμούς Θυμάστε τις φρικτές εικόνες στην τηλεόραση. Ε, σκοτώθηκαν 27 πολίτες, τραυματίστηκαν 350 πολίτες και ε, μετακινήθηκαν 45.000 πληθυσμού. Το συνολικό ποσό των ζημιών ανέρχεται σε 13 δισεκατομμύρια ευρώ. 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Θέλω να είμαι σίγουρος για αυτό που σας λέω. Αυτό σημαίνει 0,86% του Ιταλικού ΑΕΠ. Τεράστιο ποσοστό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει τέσσερις φορές το όριο το οποίο απαιτείται για να κινητοποιηθεί το συγκεκριμένο ταμείο. Ω εκ τούτου λοιπόν προτείνεται επίσημα πλέον να δοθεί μία βοήθεια 660 εκατομμυρίων ευρώ από τον προϋπολογισμό του 12 Για την κινητοποίηση αυτή λοιπόν του Ταμείου υπάρχουν κάποιες απορίες όχι. Συνεπώς μπορούμε λοιπόν να το υποβάλουμε σε ψηφοφορία αργότερα όταν έρθει η σωστή ώρα. Τώρα να έρθω στο 6. Euh, du cadre pluriannuel. Για το πολιετές πλαίσιο. Ο Ήβαλο και ο Ζων Λουκ είναι μεταξύ μας και θα με συμπληρώσουν αν χρειαστεί. Να σας παρουσιάσω πώς έχει η κατάσταση. Από την τελευταία συνεδρίαση ε, είχαμε την Τρίτη το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και χθες το πρωί συνεδρίασε η ομάδα επαφής. Ε, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και αυτό για τρίτη φορά το σύνολο της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας προσκλήθηκε σε μια ανεπίσημη συνάντηση που είχε σχέση το MFF. Ήταν στην ουσία ένα πρωινό εργασίας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 στο Λουξεμβούργο. Επί τη βάση ενός νέου λοιπόν εγγράφου εργασίας που κατέφεσε η Κυπριακή Προεδρία είναι ένα κείμενο εργασίας το οποίο ε, περιοριζόταν στην αναφορά ορισμένων οριζοντίων θεμάτων. Μακροοικονομική αιρεσιμότητα, ραλ, ευελιξία και το αποθεματικό ανάγκης και επί τη βάση του κοιτίου διαπραγμάτευσης όπως το προτείνουν οι Κύπροι, το negotiating box. Για μια ακόμη φορά λοιπόν εμείς σαν κοινοβούλιο υποδείξαμε ποια θεωρούμε κομβικά σημεία. Για να το κάνουμε αυτό φυσικά ε, στηριχθήκαμε στην ψηφοφορία της Επιτροπής Προϋπολογισμών για την ενδιάμεση έκθεση λέγοντας ότι άλλωστε το έγγραφο αυτό, το interim report, θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα. Όπως ήταν αναμενόμενο δεν υπήρξαν θεαματικά βήματα προόδου Όλοι οι υπουργοί γνωρίζουν πλέον ότι ε, οι αποφάσεις θα ληφθούν στη συγκεκριμένη περίπτωση για τις διαπραγματεύσεις από τον κύριο Βαν Ρόμπαϊ και όλοι αρκέστηκαν στο να ε, θυμίσουν τα προβλήματα και τα χαρακτηριστικά της χώρας τους. Η συζήτηση που έγινε ήταν ανάμεσα σε δύο στρατόπεδα. Από τη μία οι φίλοι αυτών που θέλουν να ξοδεύουμε καλύτερα αυτά τα οποία ε, έχουμε στη διάθεσή μας με το Ηνωμένο Βασίλειο μπροστά και από την άλλη οι φίλοι της συνοχής θα τους ονόμαζα με ηγέτη τον Σλοβάκο Υπουργό. Και αυτό γιατί ε, ξέρετε ότι η συνάντηση αυτή στο Λουξεμβούργο έγινε λίγες μέρες μετά από τη συνάντηση της Μπρατισλάβα τη συνάντηση των λεγόμενων φίλων συνοχής. Ήκοθ εννοείται ότι εμείς έχουμε εκφράσει μια γνώμη πιο κοντά σε αυτούς τη συνοχής. Αυτή είναι και η θέση του Κοινοβουλίου. Είχαμε την ικανοποίηση να διαπιστώσουμε ότι αυτό το οποίο είναι η κύρια μας μέρη από την 1η δηλαδή να μπορέσουμε να εδραιώσουμε τη διαδικασία απόφαση ε, είναι αντιληπτό από τους υπουργούς και τον πρόεδρο Φαν Ρομπάι αλλά και τους συνεργάτες του. Εδώ και πολλές εβδομάδες λοιπόν οι διαπραγματεύσεις έχουν μπορέσει να ξεκινήσουν στα πλαίσια επισήμων ή ανεπισήμων τρίμερων διαλόγων όπως ανέφεραν οι συνάδελφοι σε σχέση με το σχέδιο κανονισμού και τις πολιτικές πρέπει να χρηματοδοτηθούν από το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Προχώρα αυτή η διαπραγμάτευση με μεταβλητή ταχύτητα. Πολλές φορές το Συμβούλιο δεν είναι σε θέση να διευκρινίσει τη θέση του διότι δεν έχει ακόμα καταφέρει να επιτύχει μέσα στους κόλπους του μία συμφωνία για να παρουσιάσει ενιαία θέση εναντί του Κοινοβουλίου, αλλά οι διαπραγματεύσεις αυτές έχουν ξεκινήσει. Έχουμε συμφωνήσει θα περιμένουμε το τέλος της διαδικασίας του προϋπολογισμού για να προχωρήσουμε περισσότερο για τα στοιχεία νομικού χαρακτήρα και είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε όλα εκτός από τα αριθμητικά στοιχεία και αν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Νοεμβρίου επιτευχθεί συμφωνία για ένα κείμενο το οποίο προκαταλαμβάνει μια σειρά από αποφάσεις νομικού χαρακτήρα που πρέπει να υπόκειται στη συναπόφαση βάσει συνδίκης Λισαβόνας. Το Κοινοβούλιο δεν θα μπορέσει να δώσει τη συμφωνία του όσο δεν έχουν ληφθεί οι πρέπουσες νομικές αποφάσεις ακολουθώντας τον ουσιώδη τύπο που προβλέπουν οι συνθήκες. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημείο για το οποίο πρέπει να σας πω ότι η κατάσταση δεν είναι ιδεώδης αλλά έχουμε ως το δυνατόν περισσότερες εγγύησεις αυτή τη στιγμή. Για τους ίδιους πόρους. Εγώ αυτό το οποίο αποκόμισα από αυτή τη συνεδρία ήταν μια αισιόδοξη άποψη, ενώ ο Ζανλίκ αντίθετα μια, είχε μια απεσιόδοξη άποψη. Και τώρα μπορεί να με διορθώσει ο Ζανλίκ. Εγώ καταμετρώ το δρόμο τον οποίο έχουμε διατρέξει, ενώ ο Ζωανλή κοιτάζει το δρόμο που πρέπει ακόμα να διατρέξουμε. Αν όμως συνεκρίνουμε την κατάσταση με αυτή που ίσχυε πριν από ένα χρόνο ή ακόμα πριν από έξι μήνες για τα θέματα αυτά, ο διατρεχθής δρόμος είναι σημαντικός. Πριν όταν το εγχείρημα ουτοπικό. Ενώ τελικά το θέμα ήρθε στην ημερησία διάταξη, ο τομέας των εσόδων αναφέρεται και στο κοιτίο διαπραγματεύσεων και σε όλα τα κείμενα. Η Κυπριακή Προεδρία έχει ανακοινώσει για την επόμενη εβδομάδα ένα έγγραφο το οποίο συνοψίζει την προβληματική των ίδιων πόρων και από, τις, από τους 28 που έλαβαν το λόγο στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων η μισή τουλάχιστον αναφέρθηκαν στο θέμα αυτό. Δύο μόνο χώρε, δύο μόνο υπουργοί είπανε δεν θέλουμε ούτε να ακούσουμε για αυτό το θέμα. Επρόκειτο για τους Σουηδούς και τους Ολλανδούς. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό, κατά την απόψή μου, είναι ότι το βάρος της αποδείξεως έχει μεταφερθεί πλέον. Η ανάγκη μεταρρύθμισης του συστήματος ιδίων πόρων εδώ το βάρος αποδείξεως δεν είναι στο, στους ώμους αυτών που θέλουν να αλλάξουν το σύστημα, αλλά σε αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να το αλλάξουν και αυτή τη στιγμή δεν έχουν κανένα επιχείρημα. Εγώ έχω φυσικά το δικαίωμα άρνηση κυρία και εάν θέλετε θα το χρησιμοποιήσω. Αλλά αυτό δεν θα μας πάει μακριά. <clears throat> Είναι λοιπόν θετικά τα πράγματα. Πέραν αυτών υπάρχουν στοιχεία που είναι ο λιγότερο θετικά. Όταν πούμε εντάξει θα συζητήσουμε, υπάρχει θέληση να προχωρήσουμε. Αλλά υπάρχουν κάποιες αντιπροσωπείες χωρών που παίζουν σημαντικό ρόλο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιταλία, Γαλλία, Πολωνία, Βέλγιο, που είπαν ότι για αυτούς η τελική συμβιβαστική λύση θα πρέπει να περιλαμβάνει και τον τομέα των εσόδων, που είναι και η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλα αυτά είναι θετικά. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτή την αλλαγή νοοτροπίας χρειάστηκε ένας χρόνος. Και αν άλλαξε αυτή η αντιμετώπιση, ακόμα δεν έχουμε αρχίσει να εργαζόμαστε επί της ουσίας εκτός από το θέμα του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, για τον οποίο έχει γίνει δεκτό ότι θα υπάρχει ενισχυμένη συνεργασία. Κανείς, κανείς δεν έχει αντίρρηση στο ότι οι χώρες οι οποίες θέλουν να ε, εγκαθιδρύσουν αυτό το φόρο μέσα στα πλαίσια ενισχυμένης συνεργασίας, ότι θα μπορούν να το πράξουν. Το επόμενο ΕΚΟΦΗΝ λοιπόν μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή όπως ξέρετε χρειάζονται τουλάχιστον 9 χώρες, αλλά υπάρχουν 11 χώρες που υπέγραψαν την επιστολή πρωτοβουλίας για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η ενισχυμένη συνεργασία. Καταρχήν όμως όλες αυτές οι χώρες δεν συμφωνούν ώστε ο φόρος αυτός ακόμα και αν θεσπιστεί να τροφοδοτεί ακόμα και εν μέρη τον κοινοτικό προπολογισμό, τον ενωσιακό προπολογισμό, ιδίως η Γερμανία είναι εναντίον μιας τέτοιας ρύθμιση. Και επίση όλε αυτέ οι χώρε δεν θα συμμετάσχουν πλήρω και τρίτον, μια άλλη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχει ακόμα μελετηθεί μέχρι στιγμής. Πρόκειται για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μια θέση η οποία είναι η έκθεση Jean-Luc Dehaene, η οποία έχει εγκριθεί στην Επιτροπή μας και θα έρθει στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα. Αλλά μέχρι στιγμής το Συμβούλιο δεν έχει κάνει ούτε μία πρώτη συζήτηση για το ΦΠΑ και τους πόρους από το ΦΠΑ και μόνο επί τη βάση αυτού του εγγράφου της Προεδρίας, το οποίο προβλέπεται να δημοσιευτεί την επόμενη εβδομάδα, θα αρχίσει το Συμβούλιο να αναφέρεται στα θέματα αυτά. Μέχρι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Νοεμβρίου θα έχουμε τη συνεδρία Κορεπέρ στις 31 Οκτωβρίου και υπάρχει μοναχά ένα Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις 20 Νοεμβρίου, δύο μέρες πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με δυσκολία λοιπόν μπορεί κανείς να φανταστεί ότι μπορεί να περατωθεί μια πολιτική συμφωνία για τα έσοδα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Και κατανοώ την ε, εμβροντισία του Ζανλίκ για το θέμα αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα θέματα αυτά έχουν προχωρήσει με τρόπο ο οποίος ήταν σε κάποιο βαθμό ανέλπιστος, παρά όλα αυτά δεν είμαστε σε θέση τον Νοέμβριο να κλείσουμε την συζήτηση. Από την άλλη πλευρά. Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν όταν θέτουμε το θέμα ενός κεντρικού προϋπολογισμού για τη ζώνη του ευρώ το οποίο μας απασχόλησε την προηγούμενη εβδομάδα και δεδομένου το θέμα αυτό βρίσκεται στη μέση διάταξη του σημερινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και επομένως και του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων που έλεγε χώρα προχθές. Φυσικά αυτό ήταν ένα τμήμα στο οποίο εμεί δεν ήμασταν προσκεκλημένοι. Εγώ έθεσα αυτό το ερώτημα. Και το έθεσα αυτό το ερώτημα θέτοντας το θέμα της ενότητος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και της εκπεφρασμένης θέλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή ΣΟΥΡΕ και πιστεύω ότι οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλουν να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο αυτή την ενδιάμεση έκθεση για να τονίσουν την ανάγκη να παραμείνει ενιαίος ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υπάρχει ένα μονάχα έγγραφο το οποίο συμπεριλαμβάνει όλες τις δεσμεύσεις που έχουν να κάνουν με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και την απαραίτητη αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι μια αρχή του προπολογισμού που ισχύει σε όλες τις χώρες μας. Το ενιαίο του προϋπολογισμού είναι μια βασική δημοκρατική αρχή που επιτρέπει και τον έλεγχο της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των χρηματοδοτικών μέσων και επίσης επιτρέπει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, τον έλεγχο από τα μέσα ενημέρωσης και από την κοινή γνώμη. Και γι' αυτό το λόγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, το ΕΤΑ, να συμπεριληφθεί και πάλι στον προϋπολογισμό και ορισμένα στοιχεία τα οποία θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βγουν από τον προπολογισμό, όπω το ΙΤΕΡ, το GMS κτλ., να ξαναμπούν στον προπολογισμό με τι αντίστοιχε πιστώσει και γενικά οποιαδήποτε δέσμευση η οποία μπορεί να αναλυφθεί στα πλαίσια της Τραπεζικής Ένωσης της ενίσχυσης της ε, εποπτείας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Τραπεζικών Συστημάτων κτλ. Όλα αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν μέσα στον προπολογισμό, να δημοσιεύονται τουλάχιστον, εάν είναι διακυβερνητικού χαρακτήρα, ως παραρτήματα στον προϋπολογισμό, τα οποία δεν είναι βέβαια μέσα στο ενωσιακό πλαίσιο. Και αναφέρθηκα στο πρόβλημα το οποίο προκύπτει εάν υπάρξει ένας κεντρικός προϋπολογισμός, όπως λέγεται, για τη ζώνη του ευρώ. Τότε ο μόνος υπουργός από τους 28, γιατί και οι Κροάτες ήταν παρόντες, ο οποίος μίλησε για τον προϋπολογισμό, για τον προϋπολογισμό της ζώνης του ευρώ ήταν ο Γερμανός υπουργό, ο οποίος είπε με σαφήνεια ότι η ιδέα αυτή ερχόταν κατευθείαν από το Βερολίνο. Αλλά η λέξη προϋπολογισμός δεν ήταν η καταλληλότερη. Η πολιτική θέληση ή η ενίσχυση της αλληλεγγύης, ιδίως μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ, με τους κατάλληλους χρημα... δημοσιονομικούς ε, τρόπους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ακριβώς δημιουργία ενιαίου προπολογισμού. Στα σχέδια συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτής της εβδομάδας περιέχουν μια παράγραφο που προσέθεσε ο πρόεδρος Φαν Ρομπέι για το θέμα αυτό και δεν μιλάει πια για κεντρικό προϋπολογισμό της ζώνης του ευρώ, αλλά για fiscal capacity στα αγγλικά, δηλαδή για ικανότητες, δυνατότητες του προπολογισμού αύριο εν ώψη των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα κατανοήσουμε ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του προϋπολογισμού και των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Αλλά είναι σαφές ότι αναφέραμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα μπορούσε να δώσει συμφωνία για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο εάν δεν υπάρχουν διευκρινήσεις και σαφήνεια σε σχέση με τα σχέδια του Συμβουλίου να υπάρχουν πρόσθετοι προϋπολογισμοί, πρόσθετα κονδύλια κτλ. Οι εισηγητές μας εξάλλου προτίθενται να, να προτείνουν την ενίσχυση των αντιστοίχων παραγράφων της ενδιάμεσης έκθεσης για να τονίσουν το σημείο αυτό και έρχομαι τώρα στην συνεδρία της ομάδας επαφής που έλαβε χώρα χθες. Κατά τη διάρκεια της οποίας συνεδριάσεως, ο πρόεδρος Σούλτς ανέφερε ότι χρειαζόταν κάποιες διατυπώσεις που θα έπρεπε να μεταφέρει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και συμφωνήσαμε μαζί του για τον τρόπο με τον οποίο θα εκφράσει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δηλαδή να μεταφέρει όλα αυτά τα οποία εγώ συνοπτικά και αδέξια σας αναφέρω. Κλείσαμε λοιπόν αυτή τη συνεδρία της ομάδας επαφής προσκαλώντας τους εισηγητές να προετοιμάσουν τροπολογίες προς την ενδιάμεση έκθεση του Κοινοβουλίου οι οποίες θα μπορούσαν να κατατεθούν όχι από την Επιτροπή Προϋπολογισμών και στο όνομά της, αλλά για πολιτικούς λόγους να κατατεθούν από τις πολιτικές ομάδες, τουλάχιστον από εκείνες τις πολιτικές ομάδες που μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι μέσα σε εισαγωγικά φίλοι του δημοσιονομικού πολιετούς πλαισίου. Και έτσι αυτές οι τροπολογίες μπορούν να έρθουν στην Ολομέλεια της επόμενης εβδομάδας. Αυτά ήθελα να σας πω και ίσως ο Ήβαλο θα μπορούσε να μας πει τι ακριβώς περιεχόμενο θα έχουν αυτές τις τροπολογίες. Ναι, ναι. Και μετά βέβαια και ο Ζων Λουκ θα λάβει το λόγο, ο Ήβαλο. Ευχαριστώ πολύ. Δουλεύουμε ακόμα με τις τροπολογίες. Καθώς ο Ράιμερ έρχεται ο Πουνανά και πρέπει να ε, ολοκληρωθεί το τελικό κείμενο. Αλλά πάντως θα έχει λίγο πολύ την εξή μορφή. Καταρχάς, μία νέα αιτιολογική σκέψη που θα παραπέμπει στο άρθρο 310 της συνθήκης όπου θα λέγεται ότι κάθε δαπάνη και έσοδο ε, θα καταγράφεται στον προϋπολογισμό, κάθε δαπάνη και έσοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταγράφεται στον προϋπολογισμό. Μετά, θα υπάρχει μια άλλη αιτιολογική σκέψη η οποία θα λέει ότι ενώ ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός εξασφαλίζει εγγύηση για τις μεσοπρόθεσμες πληρωμές για τα κράτη και το EFSM επίσης εγγυάται λοιπά Δηλαδή θα υπενθυμίσουμε ότι και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός ήδη χρησιμοποιείται ή έχει χρησιμοποιηθεί για την ε, χορήγηση εγγυήσεων σε τέτοιες περιπτώσεις και τελική παράγραφος συμπεριλαμβανομένης και της διατύπωσης του κυρίου Φαν όπου θα λέμε ότι κάθε νέα δημοσιονομική δυνατότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστοχεύει στην ε, προσαρμογή σε συμμετρικές σε συμμετρικούς κραδασμούς, αυτήν η διατύπωση του κύριου Φαν Ρόμποϊ επακριβώς, θα ε, παραπέμπεται στις λειτουργίες, θα πρέπει να αναπτύσσεται μέσα στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα υπενθυμίζουμε ότι η συνθήκη προβλέπει ότι κάθε νέα δημοσιονομική δυνατότητα θα πρέπει να εγγράφεται μέσα στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου και δεδομένης μάλλον της υποχρέωσης για σεβασμό της ενότητας του προϋπολογισμού και επίσης θα ε, ζητούμε μια νέα, ένα νέο τίτλο ή κεφάλαιο στο IMF έτσι ώστε να εξασφαλίζεται διαφάνεια ορατότητα σε αυτό το τμήμα του προϋπολογισμού. Άρα είμαστε έτοιμοι να ενσωματώσουμε ένα τέτοιο νέο τίτλο στο προϋπολογισμό. Αυτές είναι οι προτάσεις μας, κάποιες μικρό προσαρμογές, τροπολογίες, γιατί υπάρχουν εξελίξεις στους ιδίου σπόρους. Ξέρετε, στην αρχή είχαμε ζητήσει να ε, συμπεριλαμβάνει τη συνεργασία για τα κρατη Τώρα όμως αυτό έχει ενσωματωθεί στις προτάσεις της Επιτροπής και έτσι δεν χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ, Βαλό. Ζων Όχι, Πρόεδρε, εγώ δεν έχω τίποτε να προσθέσω σε σχέση με τα όσα είπατε. Στην πραγματικότητα, η σημασία αυτών των προτάσεων είναι το ότι επαναφέρουμε το θέμα των ε, ιδίων πόρων και ότι ενσωματώνεται, επιζητούμε να ενσωματωθεί το EMF στον προπολογισμό για του ιδίου σχολείου, είτε δεν έχει συζητήσει καθόλου, είτε έχει συζητήσει ελάχιστα και πάντω δεν έχει συζητήσει τον ΦΠΑ. πράγμα το οποίο καταγγέλουμε στην έκθεσή μας. Για δε τον ε, φόρο των ε, συναλλαγών ήταν στο θέμα της, ε, του Hans ε, Corporation. Άλλοι θέλανε, άλλοι δεν θέλανε να το περιλάβουν τον φόρο αυτόν στους ιδίους πόρους. Ε, αυτοί που θέλαν τον περιλάβουν τον περιορίζανε μόνο στο, στο, Eurogroup. Ο κίνδυνος δηλαδή είναι στη Σύνοδο του Νοεμβρίου να έχουμε προχωρήσει σημαντικά στο MMF, αλλά, στο πολιτισμό οικονομικό πλαίσιο, αλλά για τους ιδιούς πόρους να μην έχουμε κάτι το συγκεκριμένο Ελήψη προπαρασκευής προετοιμασίας στον φάκελο αυτόν. Και φαίνεται ότι η Επιτροπή δεν είναι διατεθειμένη να καταθέσει νέε προτάσει πράγμα το οποίο θα καθίστατο το αναγκαίο, εάν δεν είναι δυνατόν αυτό ο φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών να εισαχθεί, δηλαδή αν περιοριστούμε μόνο στην πτυχή του ΦΠΑ. Πράγμα το οποίο ουσιαστικά εξηγεί και τη δική μου πρόβλεψη ότι θα βρεθούμε σε δύσκολη θέση τον Νοέμβριο έστω και αν όντω, όπως είπατε και εσείς, παραμένει επιτάπητος το θέμα. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος, για να ακολουθήσουμε λίγο και μια παρομοίωση γυναικολογική, ελπίζουμε ότι θα γεννηθεί το βρέφος, ε, φοβούμενοι όμως ότι δεν θα έχει διαστάσεις μαμούθ και κατά πόσον βέβαια θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει, να τεθεί σε λειτουργία τον Νοέμβριο όλο αυτό το οικοδόμημα. Άρα, ετοιμάζουμε τροπολογίες, καταθέτουμε τροπολογίες, παρουσιάζουμε προτροπολογίες από πλευρά των ε, πολιτικών ομάδων στις, στην Ολομέλεια. Υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις στο θέμα αυτό? Όχι, σας ευχαριστώ. Και άρα περνάμε στο προσεχές θέμα ή καλύτερα γυρνάμε στο σημείο όχι το Φερνάντες το κάναμε το 7 και θα δώσω το λόγο στη Ιούτα μία τροπολογία στον κανονισμό, μια τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή έχουμε Ιούτα ναι, Πρόεδρα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επιτήρηση εποπτείας των, το, Ευρωπαϊκός Φορέας Εποπτείας των ε, Τραπεζών ονομάζεται ε, αρχή αλλά βασικά είναι αποκεντρωμένη υπηρεσία και έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια όπως ε, διαμορφώθηκε μάλλον συγκεκριμένα με την νομοθεσία την περσινή πρέπει τώρα και επειδή οι αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων είπαν τον Ιούνιο ότι θέλουν μια ενισχυμένη επιτήρηση των τραπεζών και μόνο τότε μπορούν ε, να ε, επιτρέψουν την ε, απευθείας ανακεφαλαίωση τραπεζών από το ESF. Με αυτή την προϋπόθεση λοιπόν που όρισαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων προσπαθούμε να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Αρχή Επιτήρηση Τραπεζών και αντίστοιχα τροποποιείται ο κατάλογος των αρμοδιοτήτων της από με μια πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι θέμα νομοθεσία. Δεν έχουμε να συζητήσουμε εάν γίνεται, αν δεν γίνεται, τι έχει κάνει η Επιτροπή, τι πρέπει να τροποποιηθεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο λαμβάνει η Επιτροπή των Οικονομικών. Ω αρμόδια κατ' ουσίαν Επιτροπή, μέχρι τώρα ούτω ή άλλω δεν γνωρίζουμε τι μορφή τελικά θα πάρει αυτή η πρόταση. Αλλά σαφέ είναι ότι εμεί εδώ στη γνωμοδότησή μα με τι τέσσερι τροπολογίε ως προς τη νομική βάση, λέμε ότι θέλουμε να γνωρίζουμε από πού θα χρηματοδοτείται αυτή η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Θέλουμε να το γνωρίζουμε προκαταβολικά. Δεν θέλουμε να επιληθεί εκ των υστέρων, δηλαδή όπως έχουμε δει και στο παρελθόν, ή να δούμε μια αντιπαράθεση και διαπραγμάτευση στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση αυτής της αρχής, όπως έχει γίνει στο παρελθόν. Εφόσον λοιπόν έχει ληφθεί η απόφαση, πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας καταθέσει ένα τροποποιημένο financial sheet, ένα δημοσιονομικό δελτίο, έτσι ώστε να γνωρίζουμε τι τρέχει, τι ακριβώς συμβαίνει και έτσι επί τη βάση αυτού του νέου φάσματος του δημοσιονομικού να γνωρίζουμε εάν αυτό το οποίο σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει, αν αυτό το οποίο έχει περιλάβει δηλαδή στο σχέδιό της και στα μελλοντικά σχέδια προϋπολογισμού είναι επαρκές για τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Αυτά βέβαια και πάλι οι διαπραγματεύσεις ε, δυνάμει του άρθρου 47 με το Συμβούλιο για το πώς θα χρηματοδοτηθούν όλα αυτά. Τα έχουμε ξαναδεί, τα γνωρίζουμε. Η τρίτη τροπολογία στόχο έχει να εξασφαλίσει ότι το όποιο αποτέλεσμα ε, συναυθεί ύστερα από τα τρία χρόνια δουλειάς με το Συμβούλιο και την Επιτροπή θα υλοποιηθεί κιόλα. έχει προσδοριστεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο τα κράτη υποδοχής υπηρεσιών οφείλουν να μεριμνούν ή να προσφέρουν ε, υπηρεσίες ή κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας για τις εν λόγω υπηρεσίες. Αυτό όλο το καλύπτει η τροπολογία υπαριθμών 3. Η δε τέταρτη τροπολογία, απλά πράγματα, δεν θέλουμε η Επιτροπή να συμπεριφερθεί κατά τρόπον ώστε εκείνη να καλύψει όλη την ε, λειτουργία της ΕΜΠΑ, της Ευρωπαϊκής Τράπεζα, Αρχής Τραπεζών και να πει ότι το δικό της προσωπικό θα καλύψει τις ανάγκες κτλ. Θέλουμε να έχουμε μια σαφή εικόνα για το προσωπικό και από πού θα προέρχεται. Αυτά δημοσιονομικού χαρακτήρα λοιπόν οι παρεμβάσεις μας, οι τροπολογίες μας μέσα από την γνωμοδότηση. Θεωρητικά θα πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να είναι αυτονόητα, να μην χρειάζεται να τα πούμε. Αλλά η εμπειρία μας έχει δείξει ότι είναι καλύτερο να επισημαίνουμε ως αρχαία αρμόδια του προϋπολογισμού τα θέματα που μας αφορούν. Και αυτό ακριβώς είναι το αποτέλεσμα της επισήμανσης. Ευχαριστώ πολύ Γιούτα, ήταν ξεκάθαρο αυτό που είπες. Ερωτήσεις για τη Γιούτα, παρατηρήσεις, σχόλια, υποδείξεις. Ουχή, την ευχαριστώ. Και έτσι περνάω στο σημείο 9 με τον κύριο Σταυρακάκη. Η εισηγητή για τον Ενωσιακό Μηχανισμό πολιτική Προστασία. Παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφε. Αδελφοί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει μια πρόταση απόφαση σχετικά με τον νέο Μηχανισμό Πολιτική Προστασία τη Ένωση, προκειμένου, προκειμένου να στηρίξει, να συντονίσει και να συμπληρώσει τι δράσει των κρατών μελών στον τομέα τη πολιτική Προστασία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ο μηχανισμό Πολιτική Προστασία έχει αδιαφυσβήτητη προστιθέμενη αξία και αποτελεί μια ορατή και σημαντική έκφραση της αλληλεγγύης Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους πολίτες της, αλλά και προς τους πολίτες σε τρίτες χώρες. Η πρόταση επισκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων για την πρόληψη, την προετοιμασία και την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως γνωρίζουμε, η προετοιμασία και η πρόληψη είναι η σωστή απάντηση στις καταστροφές. Για τον λόγο αυτό, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των καταστροφών που προτείνει η επιτροπή ιδιαίτερα η έμφαση που έχει δώσει στην υποστήριξη των μεταφορών στι επιχειρήσει αντιμετώπιση των καταστροφών. δεν θα ήθελα να μπω στην διαδικασία να σα παρουσιάσω αναλυτικά κάθε τροπολογία που έχω προτείνει εξάλλου όλοι τι έχετε μπροστά στο φάκελό σα. αντί αυτού θα ήθελα να επικεντρωθώ στου δύο βασικού άξονε του σχεδίου γνωμοδότηση την αξία της πρόληψης και της συνέργειας με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης. Η πρόληψη στον τομέα της πολιτικής προστασίας είναι ύψης σημασίας, καθώς η πρόληψη των καταστροφών είναι λιγότερο κοστοβόρα από ό,τι η αντιμετώπιση τους. Θα πρέπει να διατίθενται επαρκείς πόροι στην έγκαιρη αναγνώριση των πιθανών καταστροφών, ενώ η βάση γνώσεων σχετικά με τους κινδύνους θα πρέπει να βελτιωθεί με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών. Από την άποψη αυτή, η πρόταση της Επιτροπής τα κράτη-μέλη να συντάξουν και να δημοσιεύσουν τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων μέχρι το τέλος του 2016 είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για την προσωρινή κατανομή 513 εκατομμυρίων ευρώ για δράσεις τόσο εντός όσο και εκτός Ένωση, και στο πλαίσιο του υψηλού κόστους της αντιμετώπισης καταστροφών δεν φαίνεται κύριε Πρόεδρε να είναι επαρκής για παράδειγμα στην περίπτωση των πλημμυρών που έπληξαν λιγουρία και την τοσκάνη της ιταλίας τον οκτώβριο του 2011 και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε κατοικίες επιχειρήσεις στη γεωργική δραστηριότητα και στο δίκτυο των υποδομών η συνολική άμεση ζημία όπως εκτιμάται από τις ιταλικές αρχές ανήλθε στα 722 εκατομμύρια ευρώ. Ε, ένα άλλο παράδειγμα που έλαβε χώρα στο ίδιο κράτος μέλος μέσα σε στην μόλι 7 ετών είναι η περίπτωση της κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σήμερα εξετάζομαι, δηλαδή την αλληλουχία των σεισμών που έπληξαν την περιφέρεια μίλια Ρωμάνα το Μάιο του 2012. Τα απίστευτα, το ύψο των ζημιών, το αναφέρατε ήδη κύριε Πρόεδρε ε, λίγα λεπτά νωρίτερα. Με λίγα λόγια και στις δύο περιπτώσεις τα ποσά που πρέπει να κινητοποιηθούν είναι δραματικά μεγαλύτερα από το ποσό που προτείνει η Επιτροπή για το σύνολο 7 ετών του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου για όλο τον κόσμο. Αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες εξορθολογισμού τις οποίες καταβάλουν τα περισσότερα κράτη-μέλη, η ανάγκη για συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλα χρηματοδοτικά μέσα εσωτερικών και εξωτερικών δράσεων όπως τα ταμεία που καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο και το Ταμείο Ελληνικής Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίνεται επιτακτική. Για παράδειγμα, τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη πολιτικών και παιδίσεων για την έγκαιρη αναγνώριση πιθανών καταστροφών. Στον τομέα της προληπτικής εξωτερικής δράσης θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι συνέργειες με το μέσο συνεργασίας για την ανάπτυξη και το μηχανισμό συνεργασίας στον τομέα της πυρονικής ασφάλειας Όσον αφορά την μετά την κρίση δράση, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα μεταξύ άλλων με την ανθρωπιστική βοήθεια που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με το Ευρωπαϊκό Εθελοντικό Σώμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας και με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι υπήρξαν περιπτώσεις όπου η κινητοποίησή του δεν ήταν έγκαιρη. Ω εκ τούτου, είναι σκόπιμο να επαναξετιστούν οι διατάξεις που αφορούν την κινητοποίησή του να απλουστευτούν οι κανόνες και οι διαδικασίες κινητοποίησης και να αυξηθεί η ευελιξία του. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνω την, παρουσία, την παρουσίασή μου κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σίτα. σε σχέση με αυτά που είπε ο εισηγητής μας για τη δημιουργία αυτού του νέου μηχανισμού πολιτικής προστασίας που όπως ανέφερε είναι συμπληρωματικέ δυνατότητες σε σχέση με το Ταμείο Αλληλεγγύης. Υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις. Ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ. Άλτα, Όχι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο εισηγητής ο κύριος Σταυρακάκης Νομίζω ότι το θέμα αυτό της πολιτικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών και έχω καταθέσει μια σειρά από τροπολογίες στην ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος και πιστεύω ότι σε ό,τι αφορά τα θέματα προϋπολογισμών Θα πρέπει και εδώ να υπάρξουν μέρε τροπολογίε και θα καταθέσω τροπολογίε επομένω και στην Επιτροπή μα. Συμφωνώ γενικά με αυτά που είπε ο κ. Σταυρακάκη σε σχέση με τα ταμεία και την πρότασή του. Το γεγονό ότι τα <clears throat> ταμεία αυτά πρέπει να ενισχυθούν γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκονται πολύ κάτω από το επίπεδο που είναι επαρκέ για να αντιμετωπιστούν φυσικέ καταστροφέ. Θα ήθελα όμω να πω ότι η πρόταση της Κομισιόν προτείνει ένα 53% για την πολιτική προστασία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 47% αν καταλαβαίνω σωστά τα ποσά αυτά για πολιτική προστασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την δική μου άποψη τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να τροποποιηθούν, θα πρέπει να ενισχύσουμε το τμήμα της πολιτικής προστασίας που αφορά το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μειωθεί αυτό που έχει να κάνει με το εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα απ' όλα, γιατί η χρηματοδότηση που προβλέπεται για αυτό το μηχανισμό είναι πάρα πολύ περιορισμένη καταρχήν και επίσης θεωρώ ότι είναι απόλυτα λογικό να υπάρχει ένας πραγματικός προϋπολογισμός για αυτό το εργαλείο πολιτικής προστασίας, αλλιώς δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Κάποιος άλλος θέλει να λάβει το λόγο. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον εισηγητή μας. Να υπενθυμίσω, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος, να υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι αύριο δεκάτη πρωινή ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 15 Νοεμβρίου, έτσι ώστε και η Επιτροπή Περιβάλλοντος, αρμόδια επί της ουσίας, να μπορέσει να ψηφίσει στις 28 Νοεμβρίου. Αν πάνε όλα καλά, τον Ιανουάριο θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ. Έχουμε πάει σχετικά γρήγορα στο χρονοδιάγραμμά μας. Θα περάσουμε στις ψηφοφορίες ήδη από τώρα. θα διακόψω λίγο τη συνεδρίαση για λίγα λεπτά, έτσι ώστε τα μέλη τα οποία βρίσκονται στο κτίριο αλλά όχι στην αίθουσα να μπορέσουν να έρθουν εδώ για να ψηφίσουν. Βλέπω με χαρά ότι η πολιτική ισορροπία η οποία ήταν ανύπαρκτη στην αρχή της συνεδριάσεως αποκαταστάθηκε πλέον μέσω της εξαιρετικά ποιοτική παρουσίας και ποσοτικά ιδιαίτερο σημαντικής παρουσίας της δικής μου πολιτικής ομάδας. Ανακοινώνω επίσης ότι στον ενδιάμεσο χρόνο και μιας και οι ψηφοφορίες δεν θα κρατήσουν και πάρα πολλή ώρα, να προτείνω από τώρα στους συντονιστές μετά την περάτωση της ψηφοφορίας να συνεδριάσουμε αμέσως εποφελούμενοι και από την παρουσία της διερμηνίας. Έτσι να ξεμπερδεύουμε θα έλεγα γρήγορα και να επιστρέψουμε στις εκλογικές μας περιφέρειες το ταχύτερο δυνατόν. Διακόπτω όμως τη συνεδρίαση για λίγα λεπτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξαναρχίζουμε, αλλά πρέπει να πω ότι έπαιξα σφάλμα με την διακοπή, διότι θέλοντας να διευκολύνω αυτούς που λείπανε να φτάσουν στην αίθουσα, έχασα αυτούς που ήταν μέσα, οι οποίοι αποχώρησαν. Ξέρετε ότι λέμε στα χαρλικά ότι η κόλαση είναι στρωμένη με καλές, ο δρόμος για την κόλαση μάλλον είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Εν πάση περιπτώσει μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι παρόντες όλοι, αλλά δεν βλέπω το στον των σοσιαλιστών, λέει ο πρόεδρος, θα έρθει φαντάζομαι. Πάντως νομίζω ότι μπορούν να ψηφίσουν οι πάντες δεν βλέπω να περισσεύει κανείς από καμιά ομάδα. Οι πράσινοι πάντως δεν έχουν πλεόνασμα. Ξεκάθαρα. Ε, ακολουθούμε τις ψηφοφορίες όπως προβλέπονται στην ημερήσια διάταξη και ως εκ τούτου πάμε στον διορθωτικό προϋπολογισμό υπαριθμών 4 που μας ε, ξέθεσε νωρίτερα υπαριθμών 5 διορθώνει ο μιλητή. Μας εξέθεσε νωρίτερα η Φρανσέσκα Με μια προφορική τροπολογία που σας έχει διανεμηθεί. Την ψηφίζουμε μαζί με τον διορθωτικό προϋπολογισμό και μία σημαντική διευκρίνηση ότι πρόκειται για πολιτικό για πολιτική και ε, ενδεικτική ψηφοφορία. Δεν μπορεί δηλαδή να χαρακτηριστεί νομικού χαρακτήρα. Α, να φτάνει και η κυρία Ανδρίασεν, καλώ ήρθατε στα αγγλικά. Προσπαθώ, ξέρετε, να χασομερίσω λίγο, να απασχολήσω τη συνεδρίαση μέχρι να φτάσετε κι εσείς στην αίθουσα πριν αρχίσουν οι ψηφοφορίες. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι μια ψηφοφορία για τον διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμών 5 γιατί και δεν μπορεί να είναι παρά μόνο ενδεικτική πολιτική ψηφοφορία, διότι το Συμβούλιο δεν έχει ακόμα ψηφίσει. Και εξήγησα νωρίτερα πως θέλουμε το υπαριθμόν 1 πρωτόκολλο, το προσαρτημένο συνθήκη τη Λισαβόνα, το Συμβούλιο να το ερμηνεύσει ως μια δυνατότητα για μια επιταχυμένη διαδικασία. Α, έφτασε και ο Γκόραν Φέρμε μεταξύ και άρα, επαναλαμβάνω, μπορούμε να ψηφίσουμε unblock τον διορθωτικό προπολογισμό του περιθμών. Πέντε υπέρ. Κατά. Μία ψήφος κατά, αποχές, εγκρίνεται μαζί με την προφορική τροπολογία και ευχαριστώ την Φραντσέσκα Βάλτσαρ. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου αλληλεγγύης πρόκειται για νομική βάση μόνο, έκθεση Φερνάντες υπέρ κατά αποχές αν κρίνεται. Σημείων 12 των ψηφοφοριών με τον κύριο Λάσλο Σούριαν. Τροπολογίες έχουμε? Έχουμε. Δεν είναι παρόν ο εισηγητής. Αλλά βλέπουμε σε κάθε τροπολογία. Πρόκειται και πάλι για κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου αυτή τη φορά προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. για την επιχείρηση 10 Βέστα. Δανία. Έχει αποσυρθεί η τροπολογία υπαριθμών 2, υπαριθμών 3 παρακαλώ της κυρία Τρούπελ. Είναι κατά ο εισηγητής. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Μάλιστα. Ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά, αν έχετε τις κάρτες σας. Άρα, εν τω και την ε, απαρτία μας, όλα καλά. Τι, ενδείξη, τι υπόδειξη έχουμε για την ψηφοφορία στην ομάδα μου. Α, μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καμία πίεση επί του Προέδρου. Καμία πίεση στην ασκήτη επί του Προέδρου. Πέρα τη ψηφοφορία, ψήφισαν οι πάντε για να δούμε αποτελέσματα. 12 υπέρ, 11 κατά. Ήσταν υπέρ. Et vous, vous êtes contre. Και εσείς κατά ήσασταν. Κατά ήσασταν. Ζων Λουκ. Επίσης. Άρα 13 κατά, 12 υπέρ. Α Ας ξανακάνουμε λοιπόν πρόσκλησης για να ξαναρχίσουμε. Ξανά αρχίζουμε, ξανά ψηφίζουμε την υπαριθμόν τρία τροπολογίας κατά τις οποίες στάσετε ο εισηγητής. Α ψηφίσουμε όλοι Είμαστε 25 με κάρτα παρόντες. Δουλεύουν όλες οι κάρτες. Πέρα της ψηφοφορία 12 υπέρ, 13 κατά. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ως προς τις κάρτες ψηφοφορίας, έτσι. Άρα απερίφθη. Τροπολογία 4, Πεφονσπερές, είναι υπέρ ο εισηγητής, υπέρ παρακαλώ, κατά. 2, 3. Αποχές εγκρίνεται. 5 με την ίδια συντάκτρια, ο συγκεκριτής είναι κατά. Υπέρ. Κατά. με τις ίδιες ισορροπίες νομίζω, αλλά στο ψηφίσουμε παρόλα αυτά. Υπαριθμών 5, ο εισηγητής είναι κατά της τροπολογίας, έχουν όλοι τις κάρτες τους, ψηφίσατε όλοι πέρα της ε, ψηφοφορία. 11 υπέρ, 14 κατά, απερίφθη χωρίς καμιά από εκεί. Και πάω στην τροπολογία υπαριθμών 6 του Αλεξάνδρ Άλβαρο, είναι υπέρ ο εισηγητής, υπέρ παρακαλώ, κατά. Μία ψήφος κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε μια σειρά τροπολογιών της ε, Μπερές μέχρι το τέλος της σελίδας, υπαριθμών 7, 8, 9, 10. Τέσσερις συνολικά τροπολογίες να τις δούμε. Ομού, όχι, όχι. Μάλιστα, ο κύριος Άβρο δεν θέλει. Η 7 παρακαλώ. Κατά. Κατά. Τρεις. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 8 υπέρ Κατά. Τρεις αποχές εγκρίνεται. Εννέα υπέρ. Κατά. Τέσσερις πέντε. Ε, αποχές εγκρίνεται. Η δέκα υπέρ. Κατά. Μία ψήφος. Αποχές εγκρίνεται όλες ψηφίστηκαν αλλά με διαφορετική πλειοψηφία κάθε φορά. Η 12 του κυρίου Άλβαρο είναι κατά ο εισηγητής. Υπέρ παρακαλώ. 3, 4, 5, 6, 7 κατά. Α, κατά παρακαλώ. Αποχές απερίφθη. Η 11 του κυρίου Άσχουρθ είναι κατά ο εισηγητής. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη με την διπλή ψηφία. Η 13 της κυρίας Μπερές, ο εισηγητής είναι υπέρ, υπέρ παρακαλώ κατά άποχες εγκρίνεται 14 του κύριου ο συγητής είναι κατά υπέρ παρακαλώ 4 κατά η πλειονότης αποχές απερίφθη. Η 15 της κυρίας Μπερές, ο συγητής είναι υπέρ, υπέρ παρακαλώ, κατά. Μία ψήφος κατά, αποχές εγκρίνεται. 16 των φιλελευθέρων. Ο συγκητής είναι κατά υπέρ παρακαλώ. επτά Οχτώ. Κατά. Περισσότερο από οχτώ. Αποχές ε, απερίφθη 17 της κυρίας Μπερές. Ο συγκητής είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 18 της κυρίας Μπερές. Ο εισηγητής είναι κατά αυτή τη φορά. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απερίφθη Τιολογικές σκέψεις Τροπολογία των φιλελευθέρων είναι κατά ο εισηγητής υπέρ παρακαλώ κατά Αποχές απερίφθη τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά να και είμαστε εδώ και μια και έχουμε όλες τις κάρτες γιατί όχι ψηφίζετε παρακαλώ μου λείπουν ακόμα δύο ψήφοι μία ψήφος Πέρας τη ψηφοφορία, ψήφισαν όλοι. 18 υπέρ, 4 κατά 3 αποχές και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και απουσία του. Bon, alors, euh, on, on... Λοιπόν, θα, θα την αντίστοιχη μεταφορά υπαριθμών 28 αντιστοιχεί στο πρόγραμμα το οποίο ψηφίσαμε. Η ίδια πλειοψηφία φαντάζομαι. Ποιοι είναι υπέρ, κατά. Αποχές. Γίνεται δεκτή αυτή μετά. Τώρα, κινητοποίηση του ιδίου ταμείου Για την Γερμανία όμως αυτή τη φορά, Μανρολάντ. Δεν υπάρχουν τροπολογίες εδώ. Για μια στιγμή η γραμματεία μου δεν ακολουθεί σήμερα. Τέσσερις τροπολογίες της Περβάνς. Από κοινού. Ο εισηγητής είναι υπέρ, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Τρεις είναι κατά. Αποχές και οι τέσσερις γίνονται δεκτές. Οι έξι τώρα των φιλελευθέρων, εισηγητής υπέρ Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. επτά και οκτώ της Περβόνς Μπερές. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Οι εννέα των φιλελευθέρων. Εισηγητής κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 10 της Περφάνς του εισηγητής είναι κατά ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11 και 12 μαζί. Ο εισηγητής είναι κατά και των δύο υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 των φιλελευθέρων, σε υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία η οποία είναι ηλεκτρονική. Άρχεται η ψηφοφορία. Είστε ελεύθεροι να ψηφίσετε ό,τι νομίζετε. Ο συντονιστή σας βέβαια τι λέει. Λοιπόν 18 υπέρ, 4 αποχές, 4 κατά μάλλον και 3 αποχές. Συγχαρητήρια λοιπόν. Στον εισηγητή μα. Τώρα φέτο σε ψηφοφορία και ε, την μεταφορά 27. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ιούτα και Μάρτα. Αποχές. Δεκτό. Με μια λίγο διαφορετική πλειοψηφία. Στη συνέχεια έχουμε την έκθεση Άλντα, της Άλντα, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα και έχουμε αρκετές τροπολογίες. Άλντα Σούσα. Έχουμε ένα αρκετά πλούσιο κατάλογο ψηφοφορίας. Θα μας εξηγήσει τώρα η συγγήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να πω δύο λόγια πριν από την ψηφοφορία. Καταρχήν ήθελα να πω ότι ευχαριστώ όλες τις πολιτικές ομάδες και τους εκπροσώπους τους για τη συνεργασία που είχαμε στις διάφορες συναντήσεις μεταξύ σκιωδών εισηγητών για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατό κείμενο στο θέμα αυτό. Πιστεύω ότι υπήρξε μια συνένεση και αναγνώριση της σημασίας της διατήρησης αυτού του ταμείου και φυσικά έχει υπάρξει η αίτηση να επιταχυνθούν και να απλοποιηθούν διαδικασίες οι οποίες ήταν χρονοβόρες ώστε τα άτομα τα οποία χρειάζονται την υποστήριξη από αυτό το Ταμείο να μπορούν να έχουν εγκαίρω τη χρηματοδότηση αυτή. Μετά από μια κοινή προσπάθεια που έγινε, νομίζω ότι έχουμε επιτύχει το στόχο μας. Και θα το τονίσω αυτό. Επίσης, δεν υπήρξε μια απόλυτη ομοφωνία, αλλά υπήρξε ευρεία συνένεση σε σχέση με την ανάγκη να διατηρηθεί αυτό το ταμείο μέσα στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο αλλιώς θα είχε ένα χαρακτήρα τελείως ιδεατό και πλατωνικό. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να έχει νόημα αν έπρεπε κάθε φορά να αντιμετωπίζεται χωριστά η χρήση αυτού του ταμείου. Θέλω να υπογραμμίσω ότι το ταμείο αυτό έχει ήδη βοηθήσει πάνω από 89.000 εργαζόμενους σε 20 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και χώρες των οποίων οι κυβερνήσεις είχαν αντιταχθεί στη συνέχιση αυτού του ταμείου και την προηγούμενη εβδομάδα εμείς δώσαμε κονδύλια από αυτό το ταμείο για να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους σε ορισμένες από αυτές τις χώρες που ήταν εναντίον του ταμείου. <clears throat> Θέλω λοιπόν να σας πω για τις τροπολογίες, συγκεκριμένα στην τροπολογία 53 εγώ υποστηρίζω την τροπολογία του κυρίου Κοτινή και θέλω επίσης να τονίσω δύο, ότι υπάρχουν δύο αρχικές τροπολογίες οι οποίες βρισκόντουσαν στο αρχικό κείμενο. Μία από αυτές, η τροπολογία 11, ζητά να κατέβει το κατόφλι στους 50 εργαζομένους από 200 που προβλεπόταν αρχικά και η τροπολογία 18 προτείνει να υπάρχει προσάυξηση 10% για τις χώρες σε δυσκολία και εδώ θα ήθελα και πάλι να τονίσω τη σημασία αυτής της ρήτρα. Γιατί αν σήμερα οι χώρες που έχουν προβλήματα μπορεί να είναι περιορισμένος στον αριθμό Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα προηγούμενο για το μέλλον, γιατί καμιά χώρα δεν ξέρει αν θα βρεθεί σε αντίστοιχη κατάσταση στο μέλλον και είναι χρήσιμο να υπάρχει αυτή η πρόβλεψη για μια προσάυξη 10% σε ό,τι αφορά τη βοήθεια του Ταμείου. Αυτό ευχαριστώ. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Πάμε στην λοιπόν. τώρα. Έχετε την κάρτα σας. Μάλιστα. Euh, τροπολογία 23 των φιλελευθέρων. Η συγκίτρια είναι κατά. Υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Η πλειοψηφία. Αποχές απορρίπτεται. Υπάρχει η αποκοινού ψηφοφορία για τους γεωργούς. Αν υποστηρίξετε αυτή την τροπολογία, δεν θα αναφέρεται η μνήα στους γεωργούς, αυτό θα γίνει όπου αναφέρεται η λέξη γεωργή. Είναι τρομακτικό. Αν πείτε όχι, θα αντιμετωπίσουμε τους γεωργούς. Λοιπόν, ή τους βγάζουμε τους γεωργούς ή τους βάζουμε μέσα σε όλα τα θέματα. Ποιοι είναι υπέρ της ψηφοφορίας unblock. Κατά. Δύο ψήφοι κατά. Αποχές. Πάπα λέει Γεωργή λοιπόν, τους αφαιρούμε από όλο το κείμενο όλες οι τροπολογίες και όλο το κείμενο δεν θα έχουν μνήα για τους γεωργούς. Τροπολογία 68. Το φιλελευθέρων εισηγείται είναι κατά ψήφι υπέρ. Κατά. Οι περισσότεροι απορρίπτεται. Τροπολογία συμβασμού α. Υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 73 της κυρίας Βέρτμαν. Ψήφι υπέρ. Η συγκεκριμένη είναι κατά. Κατά. Να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο παρακαλώ. Ενδιαφέρονται τα πράγματα. Και υπάρχει μια κάρτα παραπάνω από ό,τι πρέπει. Πέρας ψηφοφορίας, ελέ, εντάξει, ψηφίσατε όλοι. 15 υπέρ 11 κατά εγκρίνεται η τροπολογία αυτή. 74. Φιλελευθερών. Κατά εισηγήτρια. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Β. Συμβαστική Β. Ψήφι υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται. 11 του της συγγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική σε. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 84 εκπίπτει. Συμβιβαστική ντε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και η 88 εκπίπτει ε συμβαστική κατά αποχές δεκτή 99 Βέρτμαν η εν υπέρ ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 100 Βέρτμαν η εν κατά ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 101 Κατά εισηγητρία ψήφι υπέρ. Ναι, ναι, ναι, Κατά. Αποχές. Δεν ψήφισαν πολύ, αλλά είναι κατά οι περισσότεροι. Απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο. Αλέξανδρε. Υπάρχουν κάποιες ε, εντολές από την ομάδα του Α, υπέρ. Πολύ ωραία, πολύ Ο Αλέξανδρος έκανε μια πάρα πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση, πάρα πολύ πολύπλοκη. Και υπάρχουν ακόμα κάποιοι οποίοι δεν ξέρουν τι να ψηφίσουν. Εν πάση περιπτώσει προσπαθήσουμε να σταθμίσουμε μια θέση. Πέρασε πληροφορίες. Ψήφισαν όλοι. 12-14. Απολύτω. 102, George Lyon, η εισηγήτρια υπέρ, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, ομόφωνα. 103, της Μπάρβαρα που δεν είναι παρούσα, υπέρ, είναι και η κατά, αποχές, δεκτή. 104 κατά εισηγήτρια. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται σαφώς. 105. Είναι μια καταλανική τροπολογία από ό,τι βλέπω. Πολύ ενδιαφέρον. Η εισηγήτρια είναι υπέρ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Υποστηρίζουμε την Καταλωνία. Δεν υποστηρίζουμε τους ε, αποσχιστικούς, λέει η Γιούτα Χάουκ. είναι εσωτερικό το πρόβλημα. Δεν θα παρεμβαίναμε στα εσωτερικά του βασιλείου της Ισπανίας. 106 της Αγγέλικα Βέρτμαν. Κατά εισηγήτρια ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική F. Υπέρ. κατά αποχές υπέρ έχει εγκριθεί 109 της ε, ματέρα που είναι συμβατή ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Μπορούμε να πάρουμε τις τρεις τροπολογίες του Αλεξάνδρ Άλβαρ. Όχι. 114. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 119 Εισηγήτρια. Κατά. Ψήφι. υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 118 ματέρα, η εισηγήτρια είναι κατά. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 117 Διρό Η εισηγήτρια είναι υπέρ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 120 κοτεινή. Η εισηγήτρια είναι υπέρ. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 121-122 από κοινού, όχι, δεν μπορούμε. 121. Εισηγήτρια υπέρ, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 122. Υπέρ εισηγήτρια. εισηγειται υπερ ψηφι υπέρ, κατά. εισηγειται ψηφι υπερ δεκτή. 123 και 124 ταυτίζονται. Η εισηγήτρια το αφήνει στην κρίση της Επιτροπής. Υπέρ. ...123 και 124 υπέρ, κατά αποχές, Απολύτωνε. 125 ματέρα, η συγγήτρια δεν είναι υπέρ, ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 18 της εισηγήτριας. Συμβατή. Ναι. Η εισηγήτρια υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 130. Η συγγήτρια υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 131. Συμβαστική με την ε, συμβαστική. Υπέρ η συγκίτρια. ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 132. Εισηγητής υπέρ. Ποιος είναι υπέρ, ποι, ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή. 19. Της εισηγητρίας υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται. 133 ματέρα. Συγγήτρια υπέρ, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 134 Άλβαρο. Υπέρ η συγγήτρια, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική G. G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 139 υπέρ εισηγείται ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 138 και 140 από κοινού εισηγήτρια είναι κατά όχι δεν μπορούμε 138. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Χάνει. 100. Νομίζω ότι ψηφίσαμε την 20, λέει η κυρία Μπάλου. Έχει αποσυρθεί η 20, λέει ο Εγώ δεν έχω τροπολογία υπαριθμών 20 στον κατάλογο μου, λέει ο πρόεδρο. Έχει αποσυρθεί. Και έχασα τώρα το λογαριασμό που είμαστε. 140. Ευχαριστώ. Η εισηγήτρια κατά ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απόχε δεκτή. 141. Η εισηγήτρια είναι υπέρ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Πρέπει να κάνω έλεγχο. 141. Άρχεται η ψηφοφορία. Δύο περισσεύουνε. Δύο περισσεύουν. Έχουν βάλει την κάρτα τους, αλλά δεν ψήφισαν. Πέρα ψηφοφορίες. 15 έναντι 11 γίνεται δεκτή. 142. Εισηγητής υπέρ, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 143. Εδώ υπάρχει χωριστή ψηφοφορία, πρώτο τμήμα πρώτο τμήμα που λέει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020, η είναι υπέρ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πρώτο τμήμα της 143. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. 14-13 γίνεται δεκτό το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Είναι κατά εισηγήτρια, ψήφι υπέρ. Κατά. Ευχαριστώ, αποχές δεν γίνεται δεκτό. Περνάμε στις αιτιολογικές σκέψεις. 24 κάσα. Είναι κατά εισηγήτρια, ψήφι υπέρ. Το ΕΛΚ. Και εγώ. Κατά οι υπόλοιποι. Αποχές απορρίπτεται. Τρεις τροπολογίες της Ιζαμπέλ Τυρόμ. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί, όχι. Είκοσι Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 η συγκίτρια είναι κατά ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 Κοτίνι. η συγκίτρια είναι κατά ψήφι υπέρ κατά αποχές. Η τροπολογία αυτή λοιπόν διατηρείται, εγκρίνεται. 30. Κοτεινή εισηγήτρια υπέρ, ψήφι υπέρ, κατά. Αποχές δεκτή. 31. Καζά. Κατά εισηγήτρια, ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 των φιλελευθέρων σύγκριτρια κατά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 ματέρα σύγκριτρια υπέρ ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική H ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή 47 καζά. Ψήφι υπέρ. Η είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Η 48 είναι ταυτόσιμη. Είναι συμβατές με τι 47 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απόλυπτον οι 48 και 49. 50 Συγήτρια κατά ψήφι υπέρ. Α, εκπίπτει, με συγχωρείτε. Διότι έγινε δεκτή 47. Προφορική τροπολογία της εισηγήτριας που δεν εκπίπτει για να διαγραφεί ένα τμήμα του κειμένου. Λοιπόν, ψήφι υπέρ της προφορικής τροποποίησης της ηγήτριας. Τρει, τέσσερι, πέντε. Κατά. Η υπόλοιπη πλειοψηφία δεν γίνεται δεκτή λοιπόν. Συμβιβαστική I. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απόχες. Δεκτή. 53. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Υπέρ κατά αποχές δεκτή 54 εκπίπτει 55 η συγήτρια είναι κατά ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή 56 η συγήτρια είναι κατά ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 η εισηγήτρια είναι υπέρ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 6 και 58 είναι ταυτόσιμες. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές γίνονται δεκτές. 7 της εισηγητρίας υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε, ελέγχουμε. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά για την 7. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρασε. 12 υπέρ, 13 κατά. Και έτσι απορρίπτεται. 64 της Βαρβαρά. Η συγγήτρια είναι κατά. Υπέρ κατά αποχές απε, ε, εγκρίνεται 65 δαβητικά είναι υπέρ υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται να δούμε τις 66 και 67 μαζί όχι 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ομόφωνα 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται. Πέρας. 17 υπέρ, 4 κατά. 5 εποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια ήταν τόσο σημαντικό όσο και δύσκολο το θέμα. Και τώρα έχουμε μεταφορές ακόμα. Σημείο 15, η Φρανσέσικα παίρνει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, έχουμε ένα μεγάλο πακέτο εδώ έχουμε ήδη δύο ψηφίσει τις σχετικές με το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης την 27 και 28 αυτές τις επιστροφές λοιπόν τις ψηφίσαμε ήδη υπάρχει επίσης και μια άλλη σειρά ανάμεσά τους πιο σημαντική είναι η λεγόμενη σφαιρική δηλαδή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για όλες τις επιστροφές που μπορεί να γίνουν πριν από τον ε, προϋπολογισμό τον τροπολογι... τον νέο προϋπολογισμό τον συμπληρωματικό. Τα ποσά είναι περιορισμένα, 427 περίπου εκατομμύρια ευρώ συνολικά, ένας αριθμός ε, χαμηλότερο σχετικά με τα προηγούμενα χρόνια. Πέρυσι ήμασταν στα 700 εκατομμύρια και πριν τρία χρόνια ήμασταν στο 1 δις 700. Συνεπώς, στα πλαίσια της εφαρμογής του προϋπολογισμού, της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, έχουμε να κάνουμε με καλύτερο, θα έλεγα, αποτέλεσμα και ταυτόχρονα μας δείχνει αυτό το αποτέλεσμα ότι το μέσο αυτό των επιστροφών δεν είναι σε θέση να αλλάξει τελικά τα πράγματα παρά μόνο κατ' ολίγων. Λοιπόν, ε, έχει μείνει εκτός το 1β διότι σε αυτή την περίπτωση ε, όλα θα εξαρτηθούν από τις πληρωμές. Οι γραμμές οι οποίες θίγονται από αυτήν την επιστροφή, την σφαιρική λεγόμενη, είναι πάρα πολλές. Είναι 65 γραμμές οι οποίες ενισχύονται εκτός από, το, εκτός από τον τίτλο 1β βέβαια σε όλους τους τίτλους 45 μάλλον είναι οι γραμμές, διορθώνει η συγγήτρια. Ε, οι επιστροφές αυτές είναι όπως είπα περιορισμένες. Μόνο 13 γραμμές στον προϋπολογισμό περνούν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Πιο σημαντικό είναι το θέμα ε, της έρευνας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενισχύεται κατά 18%. 22 εκατομμύρια Γκαλιλαίο, 17 Ευρωπαϊκό ε, Δορυφορικό Πρόγραμμα Πλοήγησης. Έχουμε επίσης πάνω από 10 εκατομμύρια για τις ε, απομεμακρυσμένες περιφέρειες και την αλληλεία, την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και στον τίτλο 4, στο τμήμα 4 μάλλον, Υπάρχει επίσης ανθρωπιστική βοήθεια και 64 για την ανθρωπιστική βοήθεια και 32 εκατομμύρια για την βοήθεια σε τρόφιμα. Είπαμε 45 γραμμές, πιο σημαντικές από αυτές είναι το ίτερ 90 εκατομμύρια και μια γραμμή του προϋπολογισμού για την πυρηνική ασφάλεια, μεταβατικές δράσεις στην ουσία αποδραστηριοποίηση μονάδων παραγωγής ρεύματος, πυρηνικών μονάδων. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές γραμμές οι οποίες ωφελούνται από τις μεταφορές αυτές. Μειώνεται η βοήθεια για την ανοικοδόμηση στο Αφγανιστάν και φτάνει τα 64 εκατομμύρια Πρόκειται λοιπόν συνολικά για περιορισμένο ποσό, ένα τέταρτο αυτού που ε, επιστρέφαμε στα τέλη Οκτωβρίου πριν δύο χρόνια. Άλλες σημαντικές επιστροφές είναι οι λεγόμενες 31 και 32. Έχουμε συζητήσει για αυτές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της δημοσιονομικής για το 12 ή 31 σαν παράδειγμα αφορά την απόσυρση του αποθεματικού για το σύστημα ενημέρωσης του Σέγγεν. Είχαμε βάλει σε αποθεματικό 9 εκατομμύρια ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα κάνει κατά τη διάρκεια του 2012. Θα μας δώσει δηλαδή κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες σε σχέση με το επίπεδο προόδου του προγράμματος αυτού ενημέρωσης Schengen. Μας έδωσε τις λεπτομέρειες αυτές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε δεν τίθεται σε αυτή την περίπτωση εδώ ε, το θέμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα και το ίδιο ισχύει και για το 50% της επιφύλαξης που είχαμε βάλει για το Frontex εμείς για το 12 αφορούσε στις επιχειρήσεις της Frontex στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουν προχωρήσει και εξελίσσονται κατά τη διάρκεια του 2012 όλες αυτές οι επιχειρήσεις της Frontex, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα για να μην δοθούν τα χρήματα. Αυτά. Υπάρχουν πολύ περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά είναι περισσότερο τεχνικές ρυθμίσεις σε σχέση με την αδυναμία πληρωμών, για την αδυναμία, με την αδυναμία κινητοποίησης ταμείων κτλ. Ευχαριστώ τη Φαντσέσκα. Πράγματι λάβαμε πρόσφατα, μετά από την επεξεργασία της ημερήσιας διάταξης και μία μεταφορά υπαρίθμου 34 για τη μεταφορά 7 εκατομμυρίων ή μάλλον 0,7 εκατομμυρίων στο εσωτερικό της διαβίου κατάρτισης και αυτό θα μπορέσουμε να το ψηφίσουμε αν δεν διαφωνεί η συγγήτρια. Καλώς. Η συγγήτρια λοιπόν διευκρίνησε το περιεχόμενο από τη μία αυτού του σφαιρικού ποσού επιστροφής, αυτής της σφαιρικής μεταφοράς και από την άλλη μας ανέλησε τις επιμέρους προτάσεις μεταφοράς. Υπάρχουν διαφωνίες, ερωτήσεις, συντόνια. Ένα σχόλιο μόνο. Διαρωτώ με αν η συγγήτρια θα συμφωνήσει μαζί μου όταν διάβασα την επεξηγηματική παρουσίαση της Επιτροπής διαπίστωσα ότι πολλές από αυτές τις μεταφορές, αν όχι όλες, οφείλονται σε μορφές καθυστέρησης. Άργησε η υπογραφή της σύμβασης, οι συμμετέχοντες δεν ήταν παρόντες όταν έπρεπε κτλ. Συνεπώς, και αναφέρομαι σε γραμμές τις οποίες έχουν υπάρξει μειώσεις γενικά, περικοπές. Θα ήθελα λοιπόν να πω προς την εισηγήτρια και κυρίως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τα χρήματα αυτά τα οποία περικόπτονται τώρα ή μειώνονται τα ποσά επιστώσεις τώρα, κάποια στιγμή αργότερα σε έφετο χρόνο θα ζητηθούν πάλι, θα χρειαστούν πάλι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της συνδιαλλαγής. Δεν μιλάμε και για πάρα πολλά μεγάλα ποσά αλλά παρόλα αυτά ένα μεγάλο τμήμα αυτού του, ε, των 90 εκατομμυρίων αφορούν ε, τελικά ανάγκες οι οποίες κάποια στιγμή θα χρειαστεί να καλυφθούν και όχι πάρα πολύ μακριά μέσα στο χρόνο. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε με τις εκκρεμότητες αυτές. Γιατί επαναλαμβάνω, έχουμε να κάνουμε περισσότερο με συμβάσεις που βρίσκονται για τον ένα λόγο ή τον άλλο σε εκκρεμότητα. Και κάποια στιγμή είναι κάτι το οποίο θα επιβαρύνει το πρόβλημα πληρωμών το οποίο ήδη έχουμε σοβαρό. Φοβάμαι ότι έχετε δίκιο. Θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιδράσει πάνω σε αυτή την παρατήρηση λίγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι η σφαιρική αυτή η συνολική μεταφορά αφορά πιστώσεις πληρωμών και πρόκειται για μια ρύθμιση, κατανομή αν θέλετε, των πιστώσεων για να παρακολουθούμε κατά κάποιο τρόπο το πρόγραμμα εφαρμογής και εκτέλεσης. Συνολικά αυτό είναι το 0,3% του συνόλου των πιστώσεων πληρωμών, για να καταλάβετε το μέγεθος αν θα χρησιμοποιηθούν για εξυπηρέτηση ε, των ιδίων γραμμών στο μέλλον τα ποσά αυτά, η απάντηση είναι καταφατική. Είναι θέμα χρονοδιαγράμματος. Το θέμα είναι ότι δεν θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα ποσά τα οποία έχουν ε, ανοίξει αν θέλετε μέχρι το τέλος του χρόνου και θα χρειαστεί να τα καλύψουμε το 2013 ένα κομμάτι του τουλάχιστον μεγάλο ε, θα μεταφερθεί το 2013 με τον ένα τρόπο ή τον άλλο, θα είναι διαθέσιμα το 2013 και κατά τη διάρκεια του έτους θα υπάρχει πάντα η δυνατότητα επιμέρους ρυθμίσεων στις πληρωμές ε, μέσω ε, ενδιαμέσων πληρωμών εμβασμάτων. δεν έχουμε άλλη δυνατότητα από το να ζητήσουμε επιπλέον πιστώσεις πληρωμών μέσω ενός διορθωτικού προϋπολογισμού. Κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς για άλλους λόγους θα συμβεί την επόμενη εβδομάδα. Κοιτάξτε, τελικά το καλό νέο είναι ότι οι αξιολογήσει των αναγκών ήταν σωστές για όλες σχεδόν τις γραμμές. Το κακό νέο για μια ακόμη φορά είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τη μεταφορά αυτή παρά μόνο γιατί υπήρξαν καθυστερήσεις στις αιτήσει πιστώσεων πληρωμών. Οπότε υποχρεωτικά καλούμεθα να αυξήσουμε τις πιστώσεις πληρωμών στο μέλλον σε κάποιες γραμμές οι οποίες έτσι κι αλλιώς θα τις χαρακτήριζα ελληματικές. Και αυτό είναι κάτι, όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα συμπεριληφθεί σε έναν διαρθρωτικό προϋπολογισμό, ίσως για το τμήμα Δέλτα την επόμενη εβδομάδα και τα υπόλοιπα θα περάσουν στον προϋπολογισμό συμπληρωματικά που θα χρειαστεί να γίνει το 2013. Πάντως η εξήγηση στην παρατήρηση της συντόνια ήταν ενδιαφέρουσα και θα δούμε ακριβώς τι, ε, θα, επιπτώσεις θα έχει αυτό το φαινόμενο στο συμπληρωματικό προϋπολογισμό του 12 και στο προϋπολογισμό του 13. Λοιπόν, καλούμεθα να ψηφίσουμε αναμεταφορά. Θα ξεκινήσουμε με το 34 για, το διαβίου, για τη διαβίου κατάρτιση. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 30. Το ετήσιο συνολικό ποσό υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. 32 υπέρ. Κατά. 2 κατά αποχές 33 υπέρ κατά ένας κατά δεκτή η μεταφορά για τα άλλα τμήματα τώρα δεν έχουμε τον εισηγητή παρόντα μου είπαν ότι είναι υπέρ του συνόλου των μεταφορών, των αιτήσεων μεταφορών. Ένα πρώτο αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μια ανάγκη που έχει το δικαστήριο για τα συνταξιοδοτικά θέματα. Υπάρχουν επίσης και αιτήσει μεταφορών πάντα για το προσωπικό για το 2012. για τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής, για το λογισμικό επίσης στο 4. Εν πάση περιπτώσει έχετε τον κατάλογο νομίζω αν τον χρειάζεστε στο Κόμπου News και υπάρχει και μία επιπλέον αίτηση μεταφοράς για την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Δημοσιεύσεις και μελέτες εμπειρογνωμόνων. Σχετικά δευτερεύοντα θέματα δηλαδή. Λοιπόν, έχετε ερωτήσεις, έχετε αντιρρήσεις, μπορούμε να τα ψηφίσουμε παρακαλώ όλα μαζί αυτά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Γίνονται δεκτά. Τα αιτήματα αυτά. Λοιπόν, περνάμε τώρα στην έκθεση Αλφόνση. Α, έχει αναβληθεί η έκθεση αυτή. Τι κρίμα λέει ο πρόεδρος. Είχαμε πάρει φόρα, θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε και αυτό. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς η εισηγητής δεν είναι εδώ, αναβάλλεται. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι στα διάφορα. Α, όχι, η Γιούτα έχει κάτι στα διάφορα. Θα κάνω κάτι το οποίο θα έκανα μονάχα στην Ολομέλεια και δεν το έχω κάνει. Κάνω μια επεξήγηση ψήφου, γιατί διαπίστωσα που πολλοί εντυπωσιάστηκαν γιατί η Γιούτα Χάουκ ψήφισε κατά της κινητοποίησης του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης όπως επίσης και κατά της μεταφοράς πιστώσεων για τη Δανία και τη Γερμανία. Μα το έκανα αυτό και την τελευταία φορά εναντίον της Σουηδίας, γιατί θεωρώ ότι είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας υποχρέωσαν σε αυτήν τη ε, διαδικασία για τον προϋπολογισμό του 2012 ήταν οι οδηγές δυνάμεις για αυτή την κατάσταση και συγχρόνως έχουν την εντύπωση ότι το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης θα πρέπει να το μειώσουμε και να το σταματήσουμε στην επόμενη δημοσιονομική περίοδο και τώρα έχουν το θράσος για τα λίγα λεφτά που έχουμε να δώσουμε ως πληρωμές για τον προϋπολογισμό του 2012 να ζητήσουν να υποστηρίξουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Γι' αυτό καταψήφισε. Ευχαριστώ. Ingeborg, das haben wir letzte Mal schon besprochen. Μα τα είπαμε την άλλη φορά, Ingeborg. Βεβαίω και είναι ο προπολογισμό. Βεβαίω. Ισραίουν στον προπολογισμό τη Ευρω... της Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γερμανία. Οι εργαζόμενοι, το προσωπικό, οτιδήποτε γίνεται ή έπρεπε να έχει γίνει, έχει γίνει εδώ και καιρό ούτω ή άλλω. Και βεβαίω το Υπουργείο Εργασίας ανέλαβε δράση όπως άλλωστε πάντα συμβαίνει και δεν, δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά μόνο ότι επιτρέπουμε να ειστρέψουν τα χρήματα αυτά να επανέλθουν στον, στο γερμανικό προϋπολογισμό, στον προϋπολογισμό της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας. Αυτονόητο είναι, αλλά μου φαίνεται και αήθες το να το κάνουμε έτσι. Καλώς. Επεξήγηση ψήφου λοιπόν. Είναι... Θέλει και κύριε μια επεξήγηση. Αλλά παρακαλώ μην κολλήσουμε γιατί δεν θέλουμε τώρα να μια... Όχι, δεν είναι, δεν χρήματα πάνε στο στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία, στο Υπουργείο Οικονομικών δηλαδή, αλλά χρήματα τα οποία καταβάλλονται σε πολίτες. Δεν ε, μου φαίνεται λοιπόν σωστό το να λένε κάποιοι ότι η αλληλεγγύη ευρωπαϊκή ε, εμφανίζεται όποτε χρειάζεται. πρέπει να πηγαίνουν τα χρήματα σε αυτούς που τα χρειάζονται, όχι μόνο κατά περίπτωση. Διαφορετικά, εμείς εδώ ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχουμε βοηθήσει σε τίποτα τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και θα ήθελα να πω ότι είναι μάλλον επικίνδυνο το πεδίο στο οποίο κινείσαι. Νομίζω ότι προς φέρον όλων μας εδώ ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Εν το ήδη πόρη, λέει ο Πρόεδρος. Χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω απλώς ότι κατανοώ πλήρω τα κίνητρα που οδήγησαν τη Γιούτο Χάουκ στην στάση που παρουσίασε. Εγώ ψήφισα υπέρ και θα ψηφίσω υπέρ και για την κινητοποίηση του ταμείου αυτού σε οποιαδήποτε χώρα που κάνει μια τέτοια αίτηση γιατί θεωρώ η κρίση θα οξυνθεί, θα είναι πολύ περισσότερες χώρες οι οποίες θα χρειαστούν υποστήριξη από το Ταμείο αυτό. Καταλάβαμε ότι υπάρχει και μια σχιζοφρένεια μέσα στον πολιτικό λόγο των κυβερνήσεων που είναι κατά του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης. Είναι πράγματι κλινικού χαρακτήρα και σχιζοφρενική συμπεριφορά, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό, αλλά πιστεύω ότι το Ταμείο αυτό είναι ένα ταμείο το οποίο πρέπει να βοηθήσει τους εργαζόμενους που είναι θύματα συλλογικών απολύσεων, ανεξάρτητα από τη στάση των κυβερνήσεών τους και νομίζω ότι πρέπει να φτάσει η χρηματοδότηση του Ταμείου σε αυτούς τους εργαζομένους. Ωραία, λέει ο πρόεδρος. Εντάξει, σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήταν χρήσιμα αυτά τα σχόλια. Σας ευχαριστώ όλους. Τέλος της συνεδριάσεως. Συγχαρητήρια για την αποτελεσματικότητα όλων μας και θα ξαναβρεθούμε, οι συντονιστέ να μείνουν παρακαλώ, θα έχουμε διερμηνία στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Χρειάζεστε κάποια άλλη γλώσσα και πορτογαλικά. Ωραία, για την άλλη. Όλοι οι άλλοι διερμηνείς ελευθερώνονται. Εάν θέλουν να μείνουν, μπορούν να μείνουν μέχρι στο 10.30. Εάν όχι, κρατάμε μονάχα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και πορτογαλικά. Για δύο λεπτά διακοπή και τα ξαναλέμε στην επόμενη εβδομάδα. Πέρα στις συνεδρίες.